Uh, um, Καλημέρα σας. <clears throat> Νομίζω ότι τώρα που έχει έρθει ο εισηγητής μπορούμε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε την εξέταση της ε, ημερησίας διατάξεως που είναι εντατική γιατί είναι μίας μέρα συνεδρίαση και ε, έχουμε ε, και μέσω του διαδικτύου αναμετάδοση της συνεδριάσεως δεν ε, υπάρχουν τα νέα στοιχεία αλλά μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να βρείτε ό,τι χρειάζεστε σχετικά με την υιοθέτηση της ημερησίας διατάξεως εάν συμφωνείτε θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε ο κύριος Μπάστος ε, είναι εδώ και ανταλλάξαμε τον κύριο Ροσφόρ με την κυρία Μπάστος ε, αν λοιπόν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη σας ευχαριστώ και υπάρχουν ε, και ε, τα πρακτικά της 8ης Απριλίου και εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι το 8 το βράδυ σήμερα θα θεωρήσουμε ότι έχουν υιοθετηθεί. Τώρα λοιπόν προχωράμε σε μια σημαντική έκθεση την οποία καταρτίζει η κυρία Μπάστος για λογαριασμό μας και την χαιρετίζω διότι εντωμεταξύ ε, βλέπω ότι Αναφέρεστε στην πρόσβαση των πολιτών. Η κυρία Μπάστος λοιπόν είναι η εισηγήτριά μας και ε, πρέπει να σας πω ότι σχετικά με την ενιαία αγορά ε, πρέπει να εντοπίσουμε τις βασικές ανησυχίες ε, των πολιτών και έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση ε, από, επί του θέματος και έχουμε καλέσει διάφορες ενδιαφερόμενες ε, επί, ε, τροπές να μας στείλουν στοιχεία. Η κυρία Μπάστος επέτυχε να συγκεντρώσει στοιχεία μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός μας εφόσον εμείς εποπτεύουμε τα θέματα της ενιαίας η έκθεση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική και της δίνω το λόγο τώρα για να δούμε πώς προχωρούμε και να δούμε και τις τροπολογίες της και θα δώσω μετά το λόγο στην κυρία Μακλάκλιν ε, ε, ως εκπρόσωπο της πολιτικής μας ομάδας και αν οι σοσιαλιστές είναι εδώ επίσης θα του δώσω το λόγο. Και τώρα το δίνω στην κυρία Μπάστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα φιλικά λόγια, για τη συνεργασία μου. Το θέμα αυτό σε σχέση με τις τροπολογίες και το πώς έχει το θέμα αυτή της προκλητικής θα έλεγα έκθεσης κάποιες γενικές σκέψεις και θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην καλύτερη λειτουργία σε σχέση με τις προσδοκίες τους για τα δικαιώματά τους και την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η διάγνωση που έγινε ήταν σωστή από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν σημαντικά κενά. Ένα όσον αφορά την πληροφόρηση, ένα άλλο όσον αφορά την εφαρμογή και το νομοθετικό πεδίο. Και η δική μα στρατηγική εκπόνησης έκθεση ήταν ότι θα έπρεπε να δώσουμε προσανατολισμούς και συστάσεις και όχι τόσο απαντήσεις σε κάθε μία από τις 20 αυτές θεματολογικά υποθέσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα τρία αυτά κενά ταυτόχρονα. Έχουμε συνειδητοποιήσει πρέπει να πω εδώ και υπάρχει έντονη συνειδητοποίηση ότι αυτά τα τρία κενά θα πρέπει από καινού να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που δημιουργούν αυτά τα τρία κενά, ώστε να δράσουμε παράλληλα και συμπληρωματικά και πιθανότατα αυτές οι 20 κύριες ανησυχίες, οι κύριοι λόγοι ανησυχίες, αν δεν γίνουν αυτά, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Σε μια συγκυρία, συγκυρία κρίσης είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Εμπιστοσύνη που διακυβεύεται. Η ενιαία εσωτερική αγορά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη και επίσης για να καταφέρουμε να δώσουμε ένα μεγαλύτερο δυναμισμό, μεγαλύτερη δυναμική στις εξελίξεις και στις προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Όπως ε, είπατε Πρόεδρε, υπάρχουν διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν γνωμοδοτήσεις ε, σε σχέση με τη δική μας δουλειά αυτών των θεμάτων. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις συντάχθηκαν με βάση ένα αίτημα το οποίο είχε διατυπωθεί μέσω του Προέδρου Μάκομ Χάμπορ, ώστε σε σχέση με τις απαντήσεις ε, για αυτές τις ανησυχίες όχι τόσο ε, εξειδικευμένες προτάσεις να γίνουν, αλλά συστάσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν γενικότερα, ώστε τα κράτη-μέλη να καταφέρουν να δράσουν με το σημαντικό τους ρόλο για να μπορέσουν να επιληθούν αυτά τα θέματα. Και επίσης ε, η ανησυχία μας, ε, το μέλημά μας ήταν ε, να μην έχουμε εξειδικευμένε τοποθετήσεις, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλά από αυτά τα θέματα που αφορούν τους πολίτες έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες, ίδιες πρωτοβουλίες και με νομοθετικό έργο ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τα προσόντα, επαγγελματικά προσόντα και την δυνατότητα πρόσβασης ε, των πολιτών και σε δημόσιες ε, προμήθειες και συμβάσεις και σε σχέση με το τι γίνεται με άλλα κράτη, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο επαγγελματιών για παράδειγμα. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Όσον αφορά τις τροπολογίες τις ίδιες, κατατέθηκαν 82 τροπολογίες 24 από αυτές κατατέθηκαν από εμένα την ίδια. Και ο στόχος αυτών των 24 τροπολογιών από αυτές που κατέθεσα ήταν να εμβαθύνουμε και να ε, βελτιώσουμε το σχέδιο έκθεσης τα υπόλοιπα 58 ως προτάσεις ε, που ε, διατυπώθηκαν δεν δημιουργούν προβλήματα. Βρίσκονται στις γραμμές ε, που είχαν σκιαγραφηθεί όσον αφορά τις γενικές κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Δεν δίνουν εξειδικευμένες λύσεις για τα προβλήματα. Αυτές οι τροπολογίες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την έκθεση. Και χωρίς καμία αμφιβολία είναι βελτίωση όσον αφορά την ουσία, το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λοιπόν που κατέθεσαν τροπολογίες. Ευχαριστώ επίσης ε, συνάδελφο Ροσφόρ που κατέθεσε, Ρόμπερτ Ροσφόρ, που κατέθεσε διάφορες ε, τροπολογίες ε, που κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με τη δομή που είχε, είχαμε υπόψη για την έκθεση παρεμβαίνουν σε αυτήν και απέσυρε τις τροπολογίες 69, 71, 72, 77, 78, 79 ο κύριος Ροσφόρ. Για τις άλλες ε, τροπολογίες άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων συμφωνούμε γενικά με όλες αυτές και θα υποβάλουμε ένα σύνολο τροπολογιών, συμβιβαστικών τροπολογιών που πιστεύω ότι δεν θα δημιουργήσουν ούτε και αυτές προβλήματα στη συνέχεια δεν θα δημιουργηθούν καθόλου προβλήματα. Το αντίθετο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω δύο τροπολογίες από πλευρά του συναδέλφου Κοχέντι Κάμπου όσον αφορά το πλαίσιο τη ενιαία εσωτερική αγοράς και το κείμενο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι δύο τροπολογίες καινοτόμε πιστεύω που συνεισφέρουν με σημαντικό τρόπο για να διαμορφωθεί ε, ένα πλαίσιο επιπτώσεων όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα για τις ε, επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα μέτρα στην εσωτερική αγορά. Τέλος, Πρόεδρε, θέλω να τονίσω κάτι. Θα ήθελα να πω, να αναφερθώ στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος που ζητήθηκε για αυτό το ζήτημα, μια και πρέπει εγώ να συμμετάσχω σε μια εκστρατεία, περιφερειακή εκστρατεία στην Πορτογαλία, στη χώρα μου. Και γι' αυτό ζήτησα η συζήτηση για τις τροπολογίες να γίνει από τις 20 στις 21 Ιουνίου και η συζήτηση έτσι θα καθοριζόταν στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή στις 9 Ιουλίου. Ψήφιση στην, Κοινοβουλευτική στην Επιτροπή στις 10 και έτσι σε σχέση με τη διαβίβαση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την συνεργασία που είχα από τους συναδέλφους και συνεχίζω να αναμένω αυτή την ανταλλαγή απόψεων, προσβλέπω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όταν θα καταλήξετε θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ενσωματώσετε το ενδιαφέρον υλικό που προέρχεται από, αυτό το υλικό και γι' αυτό νομίζω ότι θα χρειαστείτε χρόνο για τις συμβιβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις διαφοροποιήσεις. Χαίρομαι που είναι τόσο εκτενείς οι παρεμβάσεις. Βλέπω ότι η κυρία Ρούλε είναι εδώ, αλλά η κυρία Μαρκλάρκ είναι η πρώτη η οποία ήταν εδώ και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε, μετά στον κύριο Σβάμπ και σε όποιο άλλο μέλος ε, θέλει, της Επιτροπής θέλει να συμμετάσχει. Η κυρία Μακλάκλιν καταρχήν. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και καλημερίζω τους δέλφους. Χαίρομαι που είναι τόσο εκτενής η έκθεση αυτή γιατί είναι μια σημαντική ανησυχία που εκφράζουν οι ψηφοφόροι μου στην περιοχή μου και πρέπει να τονιστεί, πρέπει να αντιληφθούν ότι ακούμε τις ανησυχίες τους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την έκθεση όπως η κυρία Μπάσος το ήδη είπε σήμερα το πρωί. Ε, αλλά θα εξηγήσω ορισμένα θέματα ε, που συνήθως αναφέρονται στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γι' αυτό και τονίζω τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά για να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται χρειαζόμαστε απεγνωσμένα και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διατάξεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την κατάσταση και η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της που απευθύνονται στη βιομηχανία μικρομεσών επιχειρήσεων και να αντιληφθεί ότι υπάρχει όντως ανάγκη ε, για να μειώσουν τα βάρη που ε, πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την ενιαία αγορά πρέπει να εντείνουμε τον ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου και όσον αφορά το πλαίσιο πρέπει να έχουμε έναν μηχανισμό εντοπισμού για να μπορέσουμε συγχρόνως να βελτιώσουμε και την νομική μας αγορά και ε, βέβαια οι διοικητικές πράξεις δεν είναι τόσο σημαντικές όσο οι νομοθετικές, γι' αυτό και τονίζω την πτυχή αυτή στην παράγραφο 2 και πρέπει να αξιολογήσουμε αν ε, υπάρχει προστιθέμενη αξία σε την ε, προεργασία προτού εφαρμόσουμε τις διατάξεις, να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να λαμβάνει υπόψη ε, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τους πολιτικούς και γι' αυτό θέλω να προχωρήσουμε. Γενικώ όμως ε, πιστεύω ότι πρέπει να σημειώσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες, να τις διασκεδάσουμε και προσβλέπω στη συνεργασία με την κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ κυρία Μαρκλάρκινγκ και κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά είναι κρίμα γιατί υπάρχουν ορισμένοι ευρωβουλευτές που δεν παρίστανται και ε, κάνουν τροπολογίες και θα απίφθηνα τις ε, ερωτήσεις μου σε αυτούς. Χαιρετίζω τις τροπολογίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, τις ερωτήσεις του κυρίου, της κυρίας Μπάστος. Αλλά ο κύριος Πουπάκης δεν είναι εδώ. Γιατί θέλει αυτές τις αλλαγές με την τροπολογία 13 έχω ανησυχίες και για τον κύριο Ροσφόρο. Τροπολογία 40 για το ηλεκτρονικό σύστημα. Νομίζω ότι θέλουμε να υπάρξει μία νομική βάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο και γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρωτού προβεί σε περαιτέρω διευρύνσεις να υπάρξει ε, μία έρευνα της αγοράς και αξιολόγηση και επίσης όσον αφορά την τροπολογία 65 της κυρίας Μπάστος που είναι η μοναδική ε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι εδώ αναφέρεται στο θέμα των sales law και ε, θεωρώ ότι είναι προβληματικό αν επεξεργαζόμαστε μία οδηγία και δεν έχουμε μία αποκρισταλωμένη γνώμη σχετικά με θέματα αρχής Δηλαδή αν δεν παρακολουθούμε τι γίνεται εδώ και πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν έχει επί του θέματος μία σαφή θέση. Γιατί λοιπόν σε αυτά τα θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας σε αυτό το χώρο και σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Βεβαίως εδώ έχετε ένα πολύ έγκυρο επιχείρημα, υπάρχουν θέματα που πρέπει να καλύψουμε και να που πρέπει να καλύψουμε, διότι όπως είπε η κυρία Μπάστος, πολλά από αυτά απευθύνονται στα κράτη-μέλη και ε, δεν θα έπρεπε ίσως να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η κυρία Βάιλερ τώρα και ε, νομίζω ότι μι, ε, μιλάω σαν εκπρόσωπος ενός συναδέλφου. Όχι. Όχι, δεν, δεν για τον σκιώδη Μάσα, αλλά στην ανάγνωση και του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδα κάποια θέματα τα οποία αναφύονται. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει διότι αυτά ταιριάζουν με την τελευταία παρατήρηση που έγινε το ότι εμείς δεν θα πρέπει να υπερφορτώσουμε αυτή την έκθεση με θέματα που ούτως ή άλλως είναι υπό εξέλιξη. Έχουμε και την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Όχι μόνο γνωμοδότηση, αλλά και νομοθετικό έργο κάνουμε. Όχι γνωμοδότηση για ένα πράσινο βιβλίο. Αυτό είναι το ένα που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη οι συνάδελφοι. Αν έχει νόημα να τα εντάξουμε όλα αυτά ούτω ή άλλω σε αυτό το πλαίσιο, μια και βρίσκονται ούτως ή άλλως υπό εξέλιξη νομοθετικά και από την Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος παρόν για κάποια από τα αιτιολογικά γιατί δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Γράφει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ότι το αίτιο είναι η λανθασμένη εφαρμογή κοινοτικού δικαίου. Κάπως περίεργο και απο την επιτροπη υπαρχει κάποιο παρον για καποια απο τα αιτιολογικα γιατι δεν λειτουργουν καλα τα πραγματα γραφει εδω η ευρωπαικη επιτροπη λεει οτι το βρίσκω αυτό από πλευρά της διατύπωση. Δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι ω θεματοφύλακα να μεριμνά για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αυτό είναι μια πτυχή σε αυτή τη νομοθετική, όχι νομοθετική, εκτελεστική εξουσία που δεν θα έπρεπε εμεί να επομισθούμε τέτοια καθήκοντα, αλλά να λάβουμε μόνο υπόψη με ικανοποίηση ότι έκανε σωστά τη δουλειά τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως έτσι να μα διευκολύνει. Θα μπορούσε να μα διευκολύνει αν τοποθετηθεί η Επιτροπή. Τι γίνεται με αυτή τη διατύπωση για τα κύρια πιθανά αίτια κατακαιρματισμό λέει των κεφαλαιακών αγορών ή λανθασμένη εφαρμογή κοινοτικού δικαίου. Ωραία ακούγονται αυτά, αλλά διαφορετικά αίτια τώρα, επιστροφή του φόρου, διαφορετικές εθνικές διατάξεις και ελλείψεις που υπάρχουν σε σχέση με την εφαρμογή τους. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά ίσως να μας πει κάτι η Επιτροπή περαιτέρω για να τα διευκρινίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μου υπενθυμίσατε πολύ κομψά ότι πρέπει να υποδεχθούμε τον κύριο Σονίσκι από την Επιτροπή, ο οποίο είναι εδώ και θα τον ακούσουμε μετά από ένα γύρο παρεμβάσεων των μελών. Κύριο Σουάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν εξ ονομάτων τη ομάδα του ΕΛΚ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπάστος, για την έκθεσή της και τις πολλές τροπολογίες. Τη συγχαίρω. Πιστεύω ότι η έκθεση συνολικά είναι πολύ καλή και με τα 20 σημαντικότερα θέματα των πολιτών πολύ σωστά τα λαμβάνει υπόψη αυτά τα ζητήματα στην Ευρώπη και οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, και αυτό το, το κατέδειξε η συζήτηση, τέτοιες εκθέσεις είναι κάπως γενικόλογες ή για να το διατυπώσω κάπως διαφορετικά. Είναι la langue du bois, μια ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ. Εδώ δύο θέματα αρχής θα ήθελα να τονίσω. Και αυτά που είπε η συνάδελφος Ρούιλε και η συνάδελφος Βάιλερ αφορούν κάπως το θέμα της governance, της σωστής διαχείρισης, διακυβέρνησης. Τι κάνει και πώς εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς μεριμνά και εποπτεύει για την εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη. Και τι κάνουμε εμείς ως Ευρωβουλή σε σχέση με προτάσεις που έχουν μεν συζητηθεί, αλλά σε τέτοια φυλάδια πάλι, σε τέτοιες προτάσεις πάλι αναφύονται. Η δική μου εντύπωση είναι πολλά από αυτά τα στοιχεία που αποτελούν κύρια αιτήματα των πολιτών είτε στην πράξη για την εσωτερική αγορά, είτε στην πρώτη, είτε στην δεύτερη ε, λαμβάνονται υπόψη και περιέχονται και γνωρίζουμε ότι πρέπει κάτι παραπάνω να γίνει αν δεν έχουν ρυθμιστεί, αλλά πρέπει με τη σειρά να γίνονται τα πράγματα και όχι με την αντίστροφη ε, αλληλουχία. Και όσον αφορά τα θέματα τα οποία αφορούν το υφιστάμενο δίκαιο που θα πρέπει να εφαρμόζονται, αυτό είναι το κύριο θέμα για την ενιαία εσωτερική αγορά. Δεύτερη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι η εξή. Την έκθεση την ξαναείδα άλλη μια φορά. Πρόκειται εδώ για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες, για το ψηφιακό το ψηφιακό τομέα παροχής υπηρεσιών στην, στην Ευρώπη, στην κοινοτική Ευρώπη, πανευρωπαϊκά. Ζητήθηκε για το online, για την πτυχή αυτή, να, μέσω της ε, ιστοσελίδας ε, Europe να γίνεται αυτό. Και εδώ πάλι έχουμε την αναφορά αυτής της ε, ιστοπύλης της ιστοσελίδας θα πρέπει να αποφασίσουμε και να δούμε τι θέλουμε να καταφέρουμε και δομικά να καθορίσουμε τι θα γίνεται και δεν θα επινοούμε τον τροχό κάθε μέρα εκ νέου. Είναι μια πολύ καλή έκθεση κατά τα άλλα και ευχαριστώ και για τις τροπολογίες. Ε, thank you very much. Any other... Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα μέλη τα οποία θέλουν να σχολιάσουν. Πολύ καλά. Ο κ. Βαλίνσκι μήπως θέλει να απαντήσει σε ορισμένα θέματα που εξήγησαν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μπάσες για την θαυμάσια εργασία που έκανε. Όπως είπαμε πρωτήτερα, η Επιτροπή είναι πολύ ευτυχής και χαιρετίζει το γεγονός ότι η έκθεση βρήκε σύμφωνος και ε, βεβαίως ελέγχθη πώς θα πρέπει να γίνουν ακόμα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες επιτόπου κυρίως. Δύο θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση. Πέρα από τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ορισμένα θέματα μπορεί να μην λειτουργούν στη ζωή, νομίζω ότι η Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει τα μεγαλύτερα κενά τα οποία απομένουν. Όπως εξήγησα, αυτό το κενό στην υλοποίηση δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη εφαρμογή, στο χαμηλό επίπεδο τη εφαρμογή. Προσπαθεί η Κομισιόν να καλύψει αυτό το κενό και άλλωστε έχει διαδηλώσει στο Φόρουμ τη Ενιαία Αγορά ότι μαζί με τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο 1% ε, του ελλείμματο ε, τη εφαρμογή. Παράλληλα όμω υπάρχουν άλλοι παράγοντε για του οποίου δεν λειτουργεί σωστά. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πρακτικές που ονομάζονται gold plating δηλαδή με περίπλοκες ε, ε, νομικές καταστάσεις, ε, δηλαδή αλλάζουν τις προϋποθέσεις τις καθιερωμένες. Και αυτό δεν συμβαδίζει απαραίτητα με την κοινοτική νομοθεσία και τους στόχους της. Παράλληλα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα προβλήματα αναφορά με το κενό αυτό στην εφαρμογή, η ατελής εφαρμογή των κανόνων, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και διοικήσεων και μερικές φορές τα προβλήματα έχουν σχέση με τις δυσκολίες επίλυσης αυτών και αποκατάσταση των πραγμάτων. Μερικές φορές αυτά τα πράγματα δεν αναφέρονται ε, στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Μερικές φορές χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, προκειμένου να εφαρμόζεται ο νόμος στη πράξη. Βεβαίως πρέπει να, να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και για αυτό το λόγο παρακολουθούμε συνεχώς ε, την επιτελούμενη πρόοδο. Παράλληλα όμως υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία δεν ε, μπορεί μόνη να αντιμετωπίσει η Επιτροπή. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία και συμμετοχή των κρατών μελών. Γι' αυτό με τα χαράς βλέπω ότι η έκθεση αυτή μερικές φορές στρέφεται στα κράτη-μέλη ζητώντας τους να δραστηριοποιηθούν για να μας βοηθήσουν στην υλοποίηση ε, της εσωτερική αγοράς. Θα ήθελα επίση κάτι να πω για το Europortal. Συμφωνούμε απόλυτα. Μόλι φτιάξαμε αυτή την πύλη ε, έχοντας υπόψη ένα project το οποίο θα πρέπει να είναι ενιαία σπηλή single gate για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και γι' αυτό το λόγο αναθεωρούμε συνεχώς το περιεχόμενο, προσπαθώντας να βρούμε νέους τομείς, νέους υποτομείς που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές ε, και μπορούν εύκολα να καταλάβουν τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία ορθολογισμού, ένα project ορθολογισμού, προσπαθώντας να περιορίσει τον αριθμό των ιστότοπων, εξετάζοντας ποιοι ιστότοποι ε, δεν δέχονται πολλές επισκέψεις, ε, συγκεντρώνοντας αν είναι δυνατόν, όλο το περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο. Προς το παρόν αυτά ήθελα να πω για μία ακόμη φορά ευχαριστώ για αυτό το εξαιρετικό έργο που έχετε επιτελέσει. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η σωστή προσέγγιση που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω εάν κάλυψε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν την κυρία Βάλη. Ίσως μερικά, ίσως όχι όλα. Ενώ νομίζω θα στον κύριο Μπαρνίου, ο πρόκειται να έρθει εδώ για να μιλήσει για την επόμενη σειρά συζητήσεων. Πότε θα έρθει, ρωτάει η κυρία. Θα σας πούμε. Ρώτησε η κυρία Βάιλερ. Πότε. Θα σας το πούμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δείτε στην ημέρησια διάταξη. Νομίζω ότι όσον αφορά την πύλη, την διεκτική πύλη και τι πληροφορίε, ε, νομίζω ότι είναι απόλυτα συνεπής η Επιτροπή και μπορούμε να ζητήσουμε σε μια, να έρθετε σε μια επόμενη συνάντηση, ώστε να μας δοθούν και εξωτερικές συμβουλές. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε μόνο μιας. Κυρία Μπάστος, θέλετε ίσως να συνοψίσετε πού βρισκόμαστε και τυχόν να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας και ποια είναι η συνεργασία σας με τις άλλες επιτροπές και πώς μπορούμε όλα να, να τα ενσωματώσουμε ε, σε μια συνεκτική έκθεση.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 Ε, το χρονοδιάγραμμα. Στις 10 Ιουλίου θα έχουμε την Επιτροπή και εν θα έχετε το χρόνο για να αναζητήσετε τον συμβασμό μέχρι τον Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα χρονικό κενό. Νομίζω ότι ο κ. Ροσφόρ δεν έχει φτάσει ακόμα από το Παρίσι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα καφέ μέχρι τις 10 Παρακαλώ να είσαστε ακριβώς στις 10 εδώ, διότι υπάρχει το πρόγραμμα καταναλωτών που θα χρειαστεί κάποια συζήτηση και υπάρχουν και άλλα θέματα. Γι' αυτό ανυπομονώ να σας ξαναδώ στις 10 και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Κρός θα είναι εδώ στις 3 σήμερα το απόγευμα για να μιλήσει για τα δικά της σχέδια για την ψηφιακή ατζέντα και για τα θέματα του προγράμματος της Επιτροπής της επόμενης χρονιάς. Γι' αυτό ελπίζω πολλοί από εσά να είναι εδώ και νομίζω ότι θα παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα για την κυρία Γκάλλας. Απλά ήθελα να το πω σε όλους και ελπίζω να σας δούμε και στις τρεις όλους. Λοιπόν, θα διακόψουμε για 10 λεπτά συγκεκριμένα και κατόπιν θα αρχίσουμε ακριβώς στις 10.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 Uh, Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να επανεκκινήσουμε την συνεδρίασή μας και καλωσορίζω τον κύριο Ροσφόρο που έτρεξε εδώ από το Παρίσι και ήρθε εγκαίρος ε, και σε ένα πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο για τους Γάλλους πολιτικούς και ένας πολύ ε, ενδιαφέρον μήνα, σα καλωσορίζω λοιπόν όλους και την Ζακλίν Μάινερ που είναι υπεύθυνη για τις υποθέσεις καταναλωτών στη Γενική Διεύθυνση ΙΜΚΟ και ε, ήρθε εδώ με μια ισχυρή ομάδα ε, την κυρία Μικόλ και τον κύριο Φερχόβεν χαιρετίζω τους πάντες και όσον αφορά του σκιώδης η κυρία Ρόιτοβα θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπουζουτήλ που είναι ο σκιώδης ο συγητής η κυρία Ρούιλε είναι εδώ και άλλοι ε, και εγώ θα εκπροσωπήσω την πολιτική μου ομάδα σαν σκιώδης συγητής τώρα λοιπόν Έχουμε μία, ένα σχέδιο εκτέσεως του κυρίου Ροσφόρ, ο οποίος θα το παρουσιάσει και μετά θα έχουμε τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών και θα ζητήσω από την κυρία Μάινερ να σχολιάσει και στο τέλος θα παρουσιάσουμε ε, την, ε, την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί μιλάμε για ένα σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής το οποίο ορίζει το πλαίσιο χρηματοδότησης ενεργειών ε, της Ένωσης για ε, τις πολιτικές καταναλωτών για την περίοδο 2014-2020. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι γενικά είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Επίσης συμφωνώ με τους τέσσερις στόχους που προτείνονται και που άλλωστε εντάσσονται στη συνέχεια ε, του προηγούμενου προγράμματος και θα σας πω ορισμένες λεπτομέρειες σε λίγο. Ας υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει να επιτρέψει στην Ένωση να αποκτήσει μέσα για να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση μιας ε, πολιτικής καταναλωτών που πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια εντάσσεται ε, στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και σας υπενθυμίζω μία από τι εισαγωγικέ λέξεις που υπενθύμησε η Επιτροπή στην πρότασή τη είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να μπορούν να είναι πραγματικοί παίκτε τη ενιαία αγορά. και θα ήθελα επ' αυτού να σα πω ότι ίσω εισαγωγικά δικαιολογείται το πρόγραμμα αυτό να στρέφεται περισσότερο προς το μέλλον, τονίζοντας πιο στρατηγικούς στόχους ίσως, αναφερόμενοι επίσης ε, στην ατζέντα των καταναλωτών που θα ορίσει το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής καταναλωτών για τα προσεχή έτη, μελλοντική ατζέντα. Δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε για τη μικρή δυσκολία που έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα προτού οριστικοποιηθεί η ατζέντα. Πρόκειται εδώ για ένα χρηματοοικονομικό πλαίσιο και κατανομή κονδυλίων πιστώσεων. Γνωρίζετε ότι πρόκειται ε, για ένα όχι τόσο επίβολο σχέδιο, επειδή το μέσο ποσό ετησίως ε, και κατά καναλωτήν ε, είναι 5 cents ευρώ και όχι περισσότερα. Θα θέλαμε να είχαμε περισσότερα, γνωρίζουμε παράλληλα όμως ποια είναι η δημοσιονομική μας κατάσταση. Γι' αυτό προτείνω να διατηρήσουμε τα ποσά τουλάχιστον ε, για το σύνολο του προγράμματος, ακόμα κι αν <clears throat> αναφερόμενοι ε, στην Επιτροπή, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε εν παρενθέσει μια αύξηση ε, των πόρων στο πολιετές οικονομικό πλαίσιο της τάξης του 5%. Αυτό είναι ένα σχόλιο απλά και μόνο για να επενθυμίσω τους στόχους του Κοινοβουλίου μας στα πλαίσια των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων για το σύνολο των προγραμμάτων. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω τους τέσσερις στόχους αυτού του προγράμματος. Ε, ε, ο πρώτο στόχο για μένα είναι και ο κυριότερος. Άλλωστε θα ήθελα να ενισχυθεί. Είναι εκείνο που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών στην Ευρώπη, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ, προϊόντων και υπηρεσιών που να, είναι, έχουν ασφάλεια. Γι' αυτό χρειάζεται αποτελεσματική επιτήρηση των αγορών στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπάρχει το εργαλείο APEX το οποίο πρέπει να εξυγχρονιστεί, θα πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός ε, της κοινοποίησης, της επισήμανσης των επικινδύνων προϊόντων, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση αυτών των επισημάνσεων, πε, περισσότερα από 200 για το 2010 και από αυτού προτείνω λοιπόν ο στόχος αυτός να ληφθεί υπόψη στην κατανομή ε, του προπολογισμού προς αύξηση 5% ε, από 22% σε 25%, 3% αύξηση. Αυτό είναι ο βασικός στόχος και νομίζω θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ο δεύτερος στόχος είναι ενημέρωση και εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Είναι όμως κάτι για το οποίο η αξιολόγηση των ενεργειών που ελήφθησαν στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος, όπως γνωρίζετε, δεν είναι βέβαιες. Επ' αυτού νομίζω ότι αυτός υπαριθμόν δύο στόχος, σε αυτό τον δεύτερο στόχο που αποκρίνεται στην χρηματοδότηση των μελετών και των αναλύσεων που έγιναν στην Ένωση, θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια μείωση από 37 προτείνω 34% στην κατανομή αυτού του προπολογισμού, καταρχήν επειδή η φάση ε, η πρώτη φάση έχει οριστικοποιηθεί, όλες οι πάγιες δαπάνες είναι γνωστές και θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δαπανηρών αναλύσεων και μελετών για να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αποτελεσματικές και συγκεκριμένες ενέργειες. Αναφορικά με την αξιολόγηση στον τομέα της παιδείας, Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα, είδαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις που αναγνωρίστηκαν και από την Επιτροπή. Προβλέπεται ε, να εγκαταλειφθεί υπό την παρούσα μορφή αυτό το ε, πρόγραμμα, το οποίο αντιστοιχεί ανταποκρίνεται ε, στην δικαιολόγηση της μείωσης του προπολογισμού που ανταποκρίνεται στον στόχο 2. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος Κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου άποψη, όπως είπα, η οθέτηση ε, ετησίων προγραμμάτων εργασίας αποτελούν πολιτικές επιλογές. Συνεπώς, τα όσα προτείνει η Επιτροπή, πιστεύω, δεν ανταποκρίνονται στις προνομίες που προβλέπει η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο, σε σύμφωνα με το άρθρο 290 ε, της Συνθήκης, προτείνω να δούμε πώς θα υιοθετήσουμε τα ετήσια προγράμματα ε, για να ολοκληρώσουμε επίσης τον κατάλογο των ενεργειών του παραρτήματος 1. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που ήθελα να θέσω υπόψη σας. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης υπάρχουν ορισμένε βελτιώσεις επί των δικτών κυρίως του παραρτήματος 2 σχετικά με τις προτάσεις ανά ανέφερα ήδη μερικές. Για τον στόχο υπαριθμών 2 θα ήθελα να πω ότι η υποστήριξη των οργανώσεων καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οπωσδήποτε δεν πρέπει να αναθεωρηθεί, διότι ανταποκρίνεται σε κάτι, αντιστοιχεί σε κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτές οι οργανώσεις καταναλωτών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την διάδοση των πληροφοριών, Προτείνω λοιπόν να διατηρηθεί μια μεγάλη οικονομική ισχύση αυτών των οργανώσεων καταναλωτών. Προτείνω αυτό να συζητηθεί. Επίση, δεν είναι μια καινοτομία, αλλά είναι ένα προσανατολισμό που πρέπει να αναπτυχθεί. Δηλαδή, να έχουμε ε, σημεία ιστοσελίδες που μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους, ακόμα και για τις διασυνοριακές συναλλαγές, με συγκριτικά στοιχεία για την ποιότητα, για την βιωσιμότητα κτλ. Αυτό θα μας δώσει μια μεγάλη προστιθέμενη αξία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ίσως ορισμένοι ιστότοποι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά η αξιοπιστία τους δεν είναι βέβαιη, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Ε, θα ήθελα να πω για τον τρίτο στόχο, που αφορά ε, τις δικαστικές προσφυγές, ότι πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα αυτών των μηχανισμών για επίλυση των διαφορών. Θα το αναφέρουμε αργότερα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί. Αλλά όσον αφορά το πρόγραμμα καταναλωτών, θα ήθελα να υπογραμμίσουμε έντονα το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα τα οποία... Πώς θα έλεγα... Είναι άτομα που, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα μέσα και από ε, πλευράς καλλιέργειας επίσης δεν μπορούν να, έχουν αυτά τα μέσα προσφυγής. Αυτά τα άτομα είναι με γενική ονομασία τα ευάλωτα άτομα, κυρίως τα μεγάλη ηλικία, δεν έχουν την επαρκή τεχνολογική κατάρτιση. Θα ήθελα λοιπόν γενικά να σας πω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, αυτό το θέμα της εκπαίδευσης διαβίου. Η Επιτροπή επίσης έχει υπογραμμίσει το θέμα των νέων καταναλωτών. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συμμετρία και να ληφθούν υπόψη οι διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κύκλο ζωής. Τώρα, για τον τέταρτο στόχο που αφορά το σεβασμό της νομοθεσίας, την κρίση της νομοθεσίας και των εθνικών νομοθεσιών γενικά, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή από 50-70% να περάσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, διότι πρόκειται για οργανισμούς που ε, λειτουργούν σε δίκτυο και βοηθούν πολύ τους καταναλωτές. Τόσο για θέματα διασυνοριακού χαρακτήρα, γνωρίζοντα ότι αυτά τα κέντρα θα πρέπει να γίνουν περισσότερο γνωστά, δεν είναι αρκετά γνωστά σήμερα από τους καταναλωτές. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι όσον αφορά τι γενικέ γραμμέ τη έκθεση μου και αναμένω με ανυπομονησία την, την των, ε, ε, των συναδέλφων και των σχεδόν εισηγητών για αυτές τις αναλύσεις. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Ροσφόρ γιατί θέσατε πολύ σωστά τα θέματα και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και νομίζω ότι στηρίξατε την πρόταση και νομίζω ότι η ευρεία αυτή στήριξη θα επιτρέψει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές. Έχουμε τώρα την κυρία Ιγκουάν Περές. Ε, καταρχήν όμως θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρόιτοβα, μετά την κυρία Ριγκοέν, την κυρία Ρούλε, μετά εγώ εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδας και όποιο άλλος θέλει να παρέμβει στη διάθεσή του. Η κυρία Ρόιτοβα όμως καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Α, όχι εγώ, εντάξει, συγγνώμη. Ah, thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ε, αναφερθώ σε δύο βασικά θέματα ε, τα οποία σαν ε, ε, σκιώδη συγγήτρια θεωρώ σημαντικά. Καταρχήν είναι η κατανομή πόρων και μετατόπιση από το στόχο 2 στο στόχο 1. Το ΕΛΚ πιστεύει ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να προωθηθεί το πρόγραμμα που αναφέρεται σε αυτές. Γι' αυτό και ο εισηγητής ε, προτείνει να υπάρξει ένα επιπλέον παράρτημα που να αναφέρεται σε συγκεκριμένες ε, κατανομές ε, κατά στόχο που δεν προβλεπόντουσαν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά η σκιώδη εισηγητής του ΕΛΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη του στόχου 2 με κάποιο αντιστάθισμα προς το στόχο 1 γιατί τα προϊόντα είναι πολύ σημαντικά αλλά δεν πρέπει να μειώσουμε τη χρηματοδότηση του στόχου 2 που είναι ουσιαστικά πληροφόρηση και ενημέρωση των καταναλωτών και ε, θα βοηθήσει να γνωρίζουν οι ε, καταναλωτές τα δικαιώματα δικαιώματά τους και να τα εξισκίσουν ε, υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα οποία μόνα τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια προϊόντων και ε, θα πρέπει ορισμένα να περάσουν από το δίκτυο RAPEX εξού και οι καταναλωτές πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο είναι πολύ σημαντικό σε περίοδο οικονομικής κρίσεως όπου περισσότεροι ενημερωμένοι καταναλωτές οδηγούν σε μια καλύτερη αγορά και πρέπει να δούμε ε, πόσο θα προωθήσουμε το θέμα αυτό. Οι σκιώδεις οι συγητές θεωρούν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόθεση του στόχου 2 που ε, προτείνει δράση σε συνεργασία συνεργασία με τις ε, ενώσεις καταναλωτών και γι' αυτό η σκιώδη εισήγησή μας είναι να αυξήσουμε ε, και να εντείνουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του στόχου 2 σχετικά με τα κέντρα που θα δημιουργηθούν. Ακόμη ε, και εάν υπάρξουν στοιχεία που είναι πλέον περίτα θα χρειαστεί χρηματοδότηση να ανακυκλωθεί εντός του ιδίου στόχου και να μην στραφούν, στραφεί η χρηματοδότηση αυτή σε άλλους στόχους. Επίσης χρειαζόμαστε καλής ποιότητα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα ε, για τους καταναλωτές για να μπορέσουν να προβούν σε σωστές εκτιμήσεις και επιλογές και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις προτιμήσεις και θα πρέπει να βελτιώσουμε την επεξεργασία των στοιχείων και τη σχετική δυνατότητα και να αυξήσουμε ε, την ε, συγκρισιμότητα μέσω ε, ιστοσελίδων που θα συγκρίνουν τιμές και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το θέμα αυτό βάσει των δικτών ε, και ε, στα πλαίσια ε, της συνεργασίας με, με διάφορες ομάδες. Δεν θέλουμε μόνο να εστιαστούμε σε εθνική στόχους αλλά και σε συγκρίσεις μεταξύ οργανώσεων που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και ευχαριστούμε τον ε, ε, συγητή και τους άλλους κοιόδης συγητές για την συνεργασία. Τώρα η κυρία Ιριγκόεν Περέζ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίως να ζητήσω συγγνώμη διότι έπρεπε να παρέμβω σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν μπόρεσα να ακούσω τις πρώτες πληροφορίες που μας έδωσε. Σας ζητώ συγγνώμη. Και ταυτόχρονα θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική έκθεση που συντάξατε, που ακόμα δεν είχα τον χρόνο να τη μελετήσω σε βάθος, πρέπει να πω. Αλλά θα το κάνω σύντομα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, κάποιες σκέψεις να εκθέσω. Το χαιρετίζω ότι αύξησε την πρικοδότηση κατά 5% των κονδυλίων ο εισηγητής για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις ε, όσον αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε μια εσωτερική αγορά πιο δυναμική, πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή και πιο ανταγωνιστική. Διότι πραγματικά αν θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο η κατανάλωση για την οικονομική δραστηριότητα, και έτσι πρέπει να ενισχύσουμε και να έχουμε επαρκείς πόρους και κονδύλια ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους και θα προστατεύονται και καλύτερα κατά τη διάρκεια της ζωής τους και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής όπως το υπογράμμισε ιδιαίτερα όσον αφορά τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές. Δεύτερον, συμμερίζομαι με τον εισηγητή τη σημασία που είναι μεγάλη του να ενισχύσουμε τον ρόλο των ενώσεων καταναλωτών, που πολλές φορές δεν είναι πολύ γνωστές, αλλά που διαδραματίζουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό όταν έρχεται η στιγμή να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν οι πολίτες. Και ευθυγραμμιζόμενοι με την σπανίδα των κονδυλίων είναι ε, σημαντικό να υπάρξουν πλατφόρμες για την βελτίωση της πρόσβασης στην ενημέρωση και πληροφόρηση και μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον, την εκπαίδευση και κατάρτιση των καταναλωτών. Πιστεύω ότι η προστασία των ε, ευάλωτων καταναλωτών δεν αντανακλάται, δεν ε, καλύπτεται παρκώς. Και γι' αυτό θα καταθέσω κάποιε τροπολογίε ευθυγραμμιζόμενοι με του στόχου ε, αυτή τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για του πιο ευάλωτου καταναλωτέ. Τέταρτον, ε, μένει και επιμένει ο εισηγητή για να υπάρχει πρόσβαση στα συστήματα επίλυση διαφορών ατομικών και συλλογικών. Και τέλο, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά <clears throat> για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε και τη συνεργασία που είχαμε. Και θα υπάρξει η δυνατότητα να ενισχυθούν κάποιες πτυχές με τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Ρίλε. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία και για τις εξηγήσει. Προκατέλαβε πολλές από τις ερωτήσεις μου και πιστεύω ότι στις ε, γενικές γραμμές συμφωνούμε. Έχω όμως ορισμένες ερωτήσεις και εφόσον έχουν γίνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τόσους ε, ευρωβουλευτές εγώ θα ασχοληθώ με ειδικέ ερωτήσεις σχετικά με την τροπολογία 23 στο θέμα ΟΝΤΕΡ ε, θέλω να αναρωτηθούμε εάν πρέπει να έχει κανείς διαφορετική αντιμετώπιση σε δύο διαφορετικές νομοθεσίες διότι δεν μπορεί κανείς να μετακυλεί τα θέματα σε μία άλλη νομοθεσία και να μην προχωρά στην ρύθμιση σε αυτό το νομοθετικό σχέδιο. Όσον αφορά την κυρία Ρόιτοβα στο στόχο 2 και την redirection ε, θα ήθελα να ακούσω την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλο που θεωρώ ότι δεν είναι καλή και στον συντροπολογία 44 πιστεύω ότι ουσιαστικά εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ε, αν όμως κοιτάξουμε το ηλεκτρονικό σύστημα και σε αυτό αναφερόμαστε και αν θέλουμε να το αναπτύξουμε περαιτέρω, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την προστασία δεδομένων. Δεν πρόκειται μόνο για ανταλλαγή στοιχείων αλλά και για προστασία στοιχείων και εδώ θα προβούμε σε μια σχετική τροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Ε, έχω να κάνω και εγώ ορισμένα σχόλια εν ονόματι των συναδέλφων μου και θεωρώ ότι ένα βασικό θέμα που επανακάμπτει στην Επιτροπή αυτή και έγινε τώρα η συζήτηση και με την κυρία Μπάστος σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών είναι ότι επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα και τα κράτη-μέλη επίσης ε, πέραν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς να γνωρίζουν οι πολίτες τι μηχανισμοί υπάρχουν που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Αναφέρομαι εδώ εις ε, την έλλειψη προβολής ε, των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών και πιστεύω ότι τα κέντρα αυτά τα οποία εμείς ε, επισκεπτόμαστε συχνά όπως πράξαμε και στην Κύπρο πρόσφατα παράγουν πολύ καλό υλικό χωρίς όμως να έχουν πόρους για να μπορέσουν να προβούν σε μια ευρεία ενημέρωση και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνειδητοποίηση για θέματα σημαντικά, τα eco-labels, την οικολογική σήμαση ή την ηλεκτρονική αγορά ε, που μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές για να έχουν ε, πληροφόρηση σχετικά με το τι προσφυγή μπορεί να ασκήσουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μικρή εμπλοκή των καταναλωτών καταναλωτών ε, και πρέπει να προωθήσουμε το θέμα αυτό και να <clears throat> μπλέξουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Υπάρχει επίσης ε, και ένα άλλο θέμα. Πρέπει να δούμε πόσα χρήματα επενδύουμε και πρέπει να δούμε πώς η επένδυση αυτή θα πολλαπλασιαστεί από τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια προστασίας των καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο. Και είναι θέμα επιδόσεως, διότι δεν έχουμε επαρκείς δείκτες σχετικά με την συνειδητοποίηση και την προβολή των θεμάτων των καταναλωτών και πρέπει να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους με καλύτερη συνειδητοποίηση παραδείγματος χάρη. Εάν όμως δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπλοκή των καταναλωτών, την συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων, θα πρέπει να αναλυφθούν ορισμένες δράσεις ε, σε περιοχές όπου βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ε, περιοχές όπου ορισμένοι έρχονται με τα παράπονά τους ενώ αλλού υπάρχει πολύ χαμηλότερο εμπλοκή χαμηλότερη εμπλοκή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις αγορές και με την ε, ε, συγκέντρωση και ε, να έχουμε ακριβείς στόχους για να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση και την εμπλοκή των υπηρεσιών διότι διαφορετικά αν δούμε την έκθεση της κυρίας Μπάστος όπου οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και ανησυχούν ε, για το πού πρέπει να απευθυνθούν για να επιλύσουν τα προβλήματά τους και δεν συμμετέχουν στην αγορά όπως θα έπρεπε, όλα τα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ βασικά. Ε, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις που κάνουμε σε προγράμματα για τους καταναλωτές, θα πρέπει να υπάρχει μία σημαντική ισορροπία και διασύνδεση και να υπάρξει μία εξωτερική ποιήση μέσω πληροφοριών πληροφόρησης για την αξιολόγηση, για τα κράτη-μέλη, για τις ενώσεις καταναλωτών και συγκεκριμένοι στόχοι ε, για την προώθηση ε, των στόχων αυτών, διότι για τα πράγματα που δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να ε, ενδιαφερθούν οι καταναλωτές. Και βλέπουμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα στο χώρο αυτό και οι ευάλωτοι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα προσβάσεως ε, σε ε, χώρους όπως το διαδίκτυο που απευθύνονται άλλοι και αυτοί που χρειάζονται περισσότερο αυτές τις ε, υπηρεσίες είναι αυτοί που έχουν συνειδητοποιήσει λιγότερο τις δυνατότητες αυτές και δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να υποφεληθούν. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε και σε συνδυασμό με την έκθεση της κυρίας Μπάστος, δηλαδή να συνδυάσουμε όλες αυτές ε, τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές κατά τρόπον ώστε ε, εάν δεν έχουμε ε, διαφορετικούς στόχους ε, και σπαταλάμε τις τις επενδύσεις μας αν εστιαστούμε σε έναν χώρο που μπορούν να απευθυνθούν όλοι για να λύσουν διασυνοριακά τα προβλήματά τους πράγμα που προσπαθεί να καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η που δίνεται προς αυτή την κατεύθυνση ε, θα ζητήσω από την ε, κυρία Μπάνερ να σχολιάσει αλλά προηγουμένως υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο τότε δίνω το λόγο στην κυρία Μάινερ για την έκθεση του κυρίου Ροσφόρ και για ό,τι άλλο θέμα θέλει να σχολιάσει και θα μιλήσουμε και για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις διότι είναι ε, κάτι που θέλω να σχολιάσω αλλά πρώτα ας ακούσουμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους υπαλλήλου ε, για όλη τη δουλειά που κατέβαλαν για την προετοιμασία αυτού του σχεδίου έκθεσης. Συνεργαστήκαμε πολύ θετικά όλοι μαζί και ευχαριστώ για την προσοχή που έδωσαν σε αυτό το θέμα, σε αυτή την έκθεση, σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Φυσικά με ικανοποίηση βλέπουμε ότι συνολικά από όλες τις πλευρές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής υπάρχει υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος και για την προσέγγιση του Ευρωβουλίου και της, Κοινο... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμπίπτουν και βρίσκονται πολύ κοντά οι απόψεις. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία επί των οποίων διαφωνούμε όπως θα υποθέτατε Πρόεδρε. Και εδώ δύο οριζόντια εγκάσια σημεία πρώτα που θα αναφέρω και μετά κάποιες πιο εξειδικευμένες παρατηρήσεις. Το πρώτο από αυτά είναι το θέμα των κατεντολήν πράξεων κατεξουσιοδότηση πράξεων και αυτό σε σχέση και με την επιθυμία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να διατηρούν την επιρροή τους στην χρήση των κονδυλίων αυτών. Όμως η θέση της Επιτροπής είναι σαφής και δεν είναι μια ξεχωριστή θέση για το πρόγραμμα για τους καταναλωτές, αλλά αφορά επίσης και την άποψή μας όσον αφορά όλα τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας δεν είναι μια πράξη που υλοποιεί τα κριτήρια συλλήβδην αυτών των κατεξουσιοδότησης πράξεων υπάρχουν και καθορίζον, καθορίζονται στο άρθρο 294 αρχές. Η κατεξουσιοδότηση πράξη είναι γενική, ας το πω έτσι, δράση για στοιχεία που αφορούν ε, ακροθυγός κάποια σημεία αυτού του προγράμματος και νομίζω ότι δεν ε, ικανοποιείται αυτός ο ορισμός ε, στις προϋποθέσεις του. Γι' αυτό ζητούμε να υπάρξουν κατεφαρμογή πράξεις ε, για το ετήσιο πρόγραμμα και ε, διατηρούμε αυτή μας τη θέση. Τούτου λεχθέντος όμως ε, κατανοούμε απόλυτα πρέπει να πω την επιθυμία σας να εκφράζετε τις επιθυμίες σας ε, όσον αφορά τις στοχεύσεις του ετησίου προγράμματος. Και είμαι βεβαία ότι μπορούν να εξευρεθούν συμφωνίες και ρυθμίσεις ώστε έγκαιρα να μπορούν να εκφράζονται αυτές οι απόψεις που θα εντάσσονται υστερότερα στο ετήσιο πρόγραμμα. Το δεύτερο εγκάρσιο οριζόντιο ζήτημα είναι η προτινόμενη η πρόταση για να υπάρξει ένα εξειδικευμένο πλαίσιο στο παράρτημα. Έχουμε ενδεικτική χρηματοδότηση που αφορά την ε, ε, μη ένταξη κάποιων πτυχών στον ίδιο τον κανονισμό και το ότι δεν εντάσσονται σημαίνει ότι δεν είναι μια δεσμευτική πρακτική. Αυτή είναι η ως ήθιστε διαδικασία για τέτοιου είδους προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομοθετικές και εκείνες που έχουν χρηματοδοτικούς στόχους ε, καταρχήν. Και αυτό συνάδει με το άρθρο 28 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Έγινε κατεξαίρεση αυτό. Συνήθως γίνεται αυτό όταν έχουμε συγχωνεύσεις διαφορετικών προγραμμάτων σε ένα πλαίσιο, ενιαίο πλαίσιο, ώστε να υπάρξει δυνατότητα να υπάρχει η συγχώνευση αλλά να διασφαλίζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρηματοδότησης για συγκεκριμένες δράσεις. Και σε ένα πρακτικό επίπεδο η συζήτηση σήμερα το πρωί κατέδειξε εξάλλου ότι τα κονδύλια αυτά και ο επιμερισμός τους δεν είναι ακριβής επιστήμη και θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε ποια κονδύλια θα πρέπει να κατανέμονται σε συγκεκριμένα ε, ε, συγκεκριμένη αιτήσια βάση και κατά τα άλλα διαφορετικές δράσεις μπορούν με διαφορετικό τρόπο να εξειδικεύονται. Και όπως είπε η κυρία Ρόιτοβα, αν υπάρχει μια εκστρατεία που διεξάγεται για την ασφάλεια μια συγκεκριμένη κατηγορίας προϊόντων, αυτό θα πρέπει να, κατα... να ε, εντάσσεται στην ε, ασφάλεια προϊόντων ή υπό το ε, στόχο 2, για παράδειγμα, των ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές δυνατότητες. Υπονομικό πρίσμα και πρακτικό πρίσμα δεν θα θέλαμε αυτή η ενδεικτική κατανομή να περνάει στην νομοθετική πράξη. Είναι καθαρά ενδεικτικού χαρακτήρα, έχει καθαρά ένδειξη ως στόχο μια επισήμανση. Για πιο εξειδικευμένα θέματα τώρα θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα για τους δείκτες που κάποιοι προανέφεραν στις παρεμβάσεις του ως ευρωβουλευτές. Έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα και συμμεριζόμαστε την άποψή σας ότι δεν είναι τέλειοι αυτοί οι ενδείκτες και είναι δύσκολο το εγχείρημα να βρούμε χρήσιμους και σκόπιμους δείκτες για ένα τέτοιο πρόγραμμα με τέτοια χρήση. Και σίγουρα Είμαστε με ανοιχτό ε, πνεύμα πρόθυμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας και τις ε, συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις. Όμως χρειαζόμαστε δείκτες όπου αυτό είναι εφικτό και αποτελεσματικό για το κόστος, για την συλλογή των δεδομένων. Να δούμε αν πετυχαίνουμε σωστά και σκόπιμα τους στόχους μας ή όχι αναφέρθηκε και η συνειδητοποίηση όσον αφορά τους καταναλωτές και τις ενδείξεις για διαφορετικές ε, δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, ανάπτυξη αυτών των δράσεων. Έχουμε κάποιες πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ε, εαρινή αναφορά στο scoreboard, στις επιδόσεις, ε, η τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τις απόψεις των καταναλωτών, ενώσεων καταναλωτών για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα των δράσεων και κάποια στοιχεία όσον αφορά την αξιολόγηση των αγορών ε, σε σχέση με κράτη-μέλη και δράσεις που έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, έχουμε κάποια δεδομένα ήδη αυτού του χαρακτήρα. Τώρα, τα δεδομένα τα οποία αφορούν την αναγνώριση ευρωπαϊκών υπηρεσιών ε, ευρωπαϊκών δράσεων είναι πάρα πολύ δαπανηρά να συλλεχθούν. Έχουμε κάνει τέτοιο έργο, τέτοια δουλειά ήδη κατά το παρελθόν στο survey και έχουμε την πρόθεση να επαναληφθεί αυτή η δράση μέσα σε ένα διάστημα δύο ή τριών ετών. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό ετήσια, διότι είναι πολύ δαπανηρό. Είναι ιδιαίτερα διαπανηρή διαργασία αυτή σε σχέση με, με μια δειγματοληψία ικανοποιητική ε, συλλογή τέτοιων δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι αποτελεσματική. Για τα ευρωπαϊκά κέντρα ECC σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για την ε, χρηματοδότηση. Συμφωνούμε με τα σχόλια που έγιναν ότι πρέπει να βελτιώσουμε τους συντελεστές για την αναγνώριση από πλευράς των Ευρωπαίων καταναλωτών. Έχουμε κάνει τέτοιες δράσεις το 2011 που στέφθηκαν με κάποια επιτυχία και θα θέλαμε να τα επαναλάβουμε. Όμως ε, εδώ υπάρχει το θέμα της, ε, ε, του τι γίνεται πρώτα και τι ακολουθεί, όπως η κότα και το αυγό για παράδειγμα ως ζήτημα. Εδώ, σε σχέση με την προώθηση αυτών των δικτύων, όταν υπάρχουν κονδύλια, αν όμως τα κονδύλια αυτά δειχθεί ότι δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών. Πρέπει σε με, ένα κλιμακούμενο τρόπο, βήμα προς βήμα, να ακολουθήσουμε μια διαργασία. Τώρα, οι ιστοσελίδες ε, συγκρισιμότητας ε, comparison websites sites. είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το πώς οι καταναλωτές μπορούν να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα από τις, την πληθώρα πληροφοριών με την οποία βομβαρδίζονται καθημερινά από ε, διάφορες επιχειρήσεις σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη να αναπτύσσει τέτοιου είδους ιστοσελίδες συγκρισιμότητας. Γιατί, διότι πέρα από τον ε, ιδιωτικό τομέα με ε, πρότυπα επιχειρησιακά τα οποία αναπτύσσονται και συμφωνώ με το σχόλιο ότι δεν είναι πάντα αξιόπιστα όλα αυτά και δεν είναι πάντα απόλυτα αντικειμενικά. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα τα οποία αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, όσον αφορά την δικτύωση και τι επιχειρήσεις και την δυνατότητα να υπάρχει ρυθμιστική δράση όσον αφορά τέτοιες ε, ιστοσελίδες και στοιχεία. Είναι ένα πεδίο όπου οι ενώσεις ε, καταναλωτών δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα. Εμείς θα είχαμε επιφυλάξεις να αναμειχθούμε σε τομείς όπου ήδη υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες ε, από άλλους ιδιαίτερα όσον αφορά και το, την δυνατότητα παραγωγής ε, κάποιας πρόσθετης αξίας ε, για τις οργανώσεις καταναλωτών. Ξέρουμε ότι περνούν δύσκολους καιρούς οι ενώσεις ε, καταναλωτών και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα βελτιστοποίησης των δικών τους εσόδων και πόρων. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω και νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα θέματα για την εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση. Συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγήτου ότι πρέπει να συναγάγουμε τα συμπεράσματα και να μάθουμε τα σωστά μαθήματα από την αξιολόγηση. Αντί να υπάρχει μία εκ των άνω προς τα κάτω προσέγγιση στο σχεδιασμό και εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πάμε σε μία πιο διαδραστικού χαρακτήρα εις το ε, ώστε, portal, ώστε να έχουμε την δυνατότητα ανταλλαγής των πρακτικών και να προσφέρουμε στους ε, εκπαιδευτές και τους αρμόδιους για αυτά τα θέματα να έχουν υλικό που αναπτύσσεται σε ένα κράτος μέλος με μεταφράσεις και προσαρμογές για τις εθνικές ιδιομορφίες και ανάγκες εκάστοτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προτού παρακαλέσω τον εισηγητή να απαντήσει για αυτό το θέμα ε, των ε, πράξεων και εφαρμογής των πράξεων και κατά πόσον ε, εφαρμόζονται, υλοποιούνται οι διατάξεις. Η Επιτροπή των Προέδρων έλαβε μια ενημέρωση, διότι, όπως η κυρία Μάνο γνωρίζει, δεν υπήρχε σύμνη απόψεων και από ό,τι κατάλαβα, μία από τις προτινόμενες συμφωνίες ε, είναι ένα θέμα της παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μία από τις άλλες δυνατότητες βεβαίως ε, είναι να υπάρξει ένα γενικότερο νομικό πλαίσιο στην αρχή και να, για να γνωρίζουμε πώς θέλουμε να εφαρμόζονται αυτές οι πράξεις. Ε, επικεφαλής της μονάδων μου το συζητάει, αλλά η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή το έχει υποσυζήτηση. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε με τον εισηγητή και την Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ. Είναι ένα βασικό θέμα βεβαίως. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και όχι ε, πώς θα εφαρμόσουμε τις πράξεις. Προσπαθούμε και ο πρόεδρος των ε, Επιτροπών ζήτησε της Επιτροπής ζήτησε πώς μπορούμε να έχουμε μια καθοδήγηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, ώστε το κάθε θέμα που είναι που διαπραγμάτευσε με το Συμβουλίο αναφύονται προβλήματα σχετικά ε, με τις εφαρμοστικές πράξεις. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό και υπάρχουν άλλες επιτροπές ε, που εξετάζουν ε, τις παρεμφερείς συμφωνίες και εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα είναι κατακαιρματισμένες ε, ε, προϋποθέσεις και θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά. Αυτό ήταν μια γενική παρατήρηση και θα πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο. Τώρα ο κύριος Ροσφόρ θέλει να απαντήσει στα όσα ελέγχθησαν και να συζητήσουμε και για το χρονοδιάγραμμα και άλλα θέματα. Κύριε Ροσφόρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσουν μια συζήτηση λεπτομερή με τις ε, πράξεις εφαρμογής ή πράξη χωρίσεως είναι οριζόντιο θέμα και αφορά πολλές επιτροπές παρά το γεγονός ότι είμαστε μεταξύ των πρώτων επιτροπών που βλέπει αυτό το θέμα κατάματα αν θέλετε και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή τοποθέτηση μεταξύ όλων των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει επίσης να προασπίσουμε τις θέσεις μας με σαφήνεια. Αναφορικά με τα διάφορα θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα οι σκιώδει εισηγητέ. Για την κυρία Ρότοβα και θα ήθελα να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που υποστήριξε την πρότασή μου ε, για τις ε, εκχωρούμενες πράξεις. Αυτά τα θέματα τα αντιλαμβάνουμε, τα ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, όσον αφορά το switch που αφορά την οικονομική κατανομή μεταξύ των τεσσάρων στόχων. Θα ήθελα να σα πω ότι αυτή η κατανομή δεν αμφισβητεί το γεγονό ότι η παριθμόν 2 στόχο είναι ο πιο σημαντικό, επειδή με 34% ε, παραμένει ο κύριος στόχος σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα όμως, αυτή η αλλαγή του 3% από το στόχο 1 προς το 2 ε, σημαίνει συγχρόνως ότι ε, στα πλαίσια παγκοσμιοποίησης που αφορά τις πρακτικές κατανάλωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας. Για τα προϊόντα της, τα κινέζικα υπάρχουν ε, πολλά προϊόντα στις 15, το 15% των περιπτώσεων όπου δεν μπορούμε να βρούμε ποια είναι η εταιρεία που παρήγαγε αυτά τα προϊόντα. Αυτά αφορούν και το ρουχισμό αλλά και τα παιχνίδια. Πολύ σημαντική τομή για τα παιδιά μας και για τα παιδιά ε, μέσα στα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της Ευρώπης. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Δεύτερον, σχετικά με το δεύτερο στόχο, αυτή η μικρή μείωση, νομίζω, οφείλεται στο γεγονός επίσης ότι πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί, πιο αποτελεσματικοί, πιο λειτουργικοί ως προς αυτούς τους δείκτες. Το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αρμπόρος, σκιώδης εισηγητής ε, της ομάδας σας, ας μη συγχαίουμε τις αρμοδιότητες, δεν πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτοί οι δείκτες. Θα πρέπει για να μπορούν οι καταναλωτές να βρουν το δρόμο τους, θα πρέπει αυτή η δίκτης να είναι σαφής και θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε ε, τη μόχλευση με τα κράτη-μέλη. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την τοποθέτηση. Η κυρία Ριγκογιάν μίλησε για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Στην έκθεσή μου ε, προτείνω να λάβουμε υπόψη τη θέση του, την ουσιαστική του θέση όσον αφορά τι δικαστικέ προσφυγές. Αλλά η κυρία θα κάνει προτάσεις βελτίωσης του κειμένου για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές και σε άλλους τομείς και βεβαίω θα τους εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Τώρα θα ήθελα να πω στην κυρία Ρούλε ότι αναφορικά με την τροπολογία 23 αυτό έχει σχέση με τα όσα είπα για τους δείκτες, με τα όσα είπε ο ότι ο στόχος μας, όταν μιλάμε για τις ODR και ODR είναι να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή καλών πρακτικών, δηλαδή ε, να ε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, χρησιμοποιώντας, βέλτιστοποιώντας τις θετικές μας εμπειρίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Κυρία Ρούλε, επίσης, μίλησε για την τροπολογία 44. Αυτή η τροπολογία 44 πράγματι αφορά τον εξυγχρονισμό ε, των εργαλείων πληροφόρησης και πληροφορικής και των βάσεων δεδομένων. Διευκρινίζω ότι δεν μιλάμε για επεξεργασία μεμονωμένων δεδομένων, αλλά δεδομένων που αφορούν υπάρχοντα συστήματα σχετικά με τις οικονομικ... ανταλλαγές οικονομικών στοιχείων και καταναλωτικών στοιχείων. Συνεπώς δεν απειλούνται τα μεμονωμένα άτομα εδώ. Αλλά βεβαίως συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να εξακριβώσουμε ή μάλλον να ενισχύσουμε ε, την επικύρωση αυτών των δεδομένων. Τώρα, για την Επιτροπή, για την Κομισιόν, θα ήθελα, ή μάλλον συζητήσαμε ήδη για την εκχώρηση των πράξεων Τώρα, για την κατανομή των κονδυλίων του προπολογισμού. Καταλαβαίνω πολύ καλά την άποψη της Κομισιόν, η οποία λέει ότι είμαστε συμπαθητικοί μαζί σας, πολύ καλοί, σας δίνουμε αυτή την ε, κατανομή και εσείς τελικά τι θέλετε, θέλετε να γίνει μια οδηγία υπό την έννοια ότι θέλετε να, να τροποποιηθεί αυτή η κατανομή. Το καταλάβαμε αυτό. Λοιπόν, η κατανομή που προτείνουμε εμείς Εκτό από την εξαίρεση μεταξύ των προγραμμάτων 1 και 2, είναι η ίδια η κατανομή που προτείνετε εσεί. Συνεπώς συμφωνούμε με εσά. Και είδατε ότι υπάρχει και το στοιχείο της ευελιξίας είναι πλήν 20% και εδώ διευκρινίζω ότι πρέπει να το δούμε οριζόντια το θέμα, διότι σε άλλα προγράμματα γίνεται η ίδια συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής για την κατανομή των κονδυλίων. Τέλος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι το γνωρίζετε πλέον, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών έχει οριστεί στις 14 Μαΐου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Και κατόπιν θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 20 Ιουνίου, ε, στην Ολομέλεια, το 20 Ιουνίου 2012. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος και όλων των σχεδόν εισηγητών προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση αυτής της ικανοποιητικής συμφωνίας, διότι είναι καταλητική σημασία για το έργο που επιτελούμε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία μάντα που, μας, που ήρθε εδώ σήμερα το πρωί. Τώρα θα έρθουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα όσον αφορά την ενιαία αγορά για τα προϊόντα τον κανονισμό εναρμόνισης του επίπεδου ήχου και έχει πολύ για τα μηχανήματα και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το επίπεδο ηχοστάθμη δηλαδή των μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτό πρέπει να ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο, να δούμε ποια οχήματα είναι υπεύθυνα για την αύξηση της ηχοστάθμης και επίση πρέπει να έχουμε μια συνοχή εδώ, συνεκτική αντιμετώπιση όσον αφορά την ηχοστάθμη για τα μηχανοκίνητα οχήματα συγκεκριμένα. Η κυρία Βάις έκανε μια πολύ λεπτομερή δουλειά εδώ. Επίσης υπάρχει η κυρία Βέστφαλ που είναι σκιώδης ηγητής, ο κύριος Μάντες, ο οποίος είναι εδώ, κύριε Ρούλερ, και εγώ είμαι σκιώδης ηγητής για τη δική μου την ομάδα Λοιπόν, είναι η πρώτη ευκαιρία να γίνει συζήτηση του θέματος και κατόπιν έχουμε κάποιον από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ναι, κάποιος είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Πολύ καλά. Αργότερα θα σας καλέσω. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της και μετά θα γίνει ένας γύρος παρεμβάσεων από τους φιόδους εισηγητές και θα καλέσω κατόπιν την Επιτροπή να απαντήσει. Η κυρία Βάις Γκέρμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Μάκομ Χάρμπερ. Αξιότιμοι σκιώδεις εισηγητές, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής είχαμε την πρώτη ευκαιρία ανταλλαγών απόψεων για αυτό το χαρτοφυλάκιο από την αρμόδια για το θέμα Επιτροπή έχουμε και το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας πρότειναν ή μας επέβαλαν τον Ιούλιο θέλουν να ψηφίσουν και είναι σημαντικό εμείς πιο πριν να συντονιστούμε χρονικά με τη γνωμοδότησή μας ώστε να ληφθεί έγκαιρα υπόψη και γι' αυτό τον λόγο κατέθεσα και την έκθεσή μου την οποία ξεπώνησα την τελευταία φορά και άμεσα στα αγγλικά σας την διαβίβασα τώρα είναι διαθέσιμη στις διάφορες γλώσσες και είχαν την ευκαιρία να, οι συνάδελφοι να δουν αυτά τα θέματα, οι οι εισηγητές, ε, τα πιο σημαντικά θέματα πρώτα, γενικά. Είναι ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο για την προστασία της υγείας. Πάλι ένα θέμα που αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα, όχι όμως τις βλαπτικές ουσίες και τις εκπομπές ρήπων, αλλά την ηχοστάθμη της ηχορύπανσης. Όσον αφορά τα ΙΧ και τα φορτηγά πρέπει να γίνουν πιο λιγότερο ηχητικά ενοχλητικά με μικρότερη εκπομπή ρήπων. Ο θόρυβος ε, δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορικά, ε, καρδιακά, του ύπνου ή ακόμα και της, ε, του συντονισμού και υπάρχουν συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πόσοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τακτά διαστήματα εκτίθενται σε τέτοιου είδους χορύπανση και ηχητική όχληση. Πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα όπως και με την ποιότητα της ατμόσφαιρας και του αέρα που αναπνέουμε για την προστασία της υγείας των καταναλωτών να μειωθεί η χορύθμα, η Τώρα για τη γνωμοδότησή μου. Προσπάθησα στη γνωμοδότησή μου να επικεντρωθώ σε αυτά τα θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Αυτό το θέμα θέλω κυριότερα να θέσω στο επίκεντρο. Πληροφορίες για τους καταναλωτές λοιπόν. Θα χαιρόμουν αν σε αυτό το σημείο καταλήγαμε σε μια κοινή τροπολογία που θα υιοθετούσαμε διακομματικά και αυτή την εβδομάδα έχουμε μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών που έχει προβλεφθεί για να σφιγμομετρήσουμε τα πράγματα, να δούμε ποιε είναι οι απόψει και με του συναδέφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε συζητήσει που ήταν, υπήρχε ανοιχτή, ε, ανοιχτό πνεύμα για, και από πλευρά των σοσιαλδημοκρατών και για την ετικετοποίηση και επισήμανση για το labeling. Έχουμε τέτοιου είδου ε, labeling για τι ε, εκπομπέ ρήπων αλλά και επίση και για τους, την ηχητική ρήπανση που προκαλείται από τα λάστιχα Υπάρχει λοιπόν πρόθεση, μια και υπάρχει ήδη πείρα σε αυτό τον τομέα, να προχωρήσουμε. Και οι εκπομπές ρήπων ε, για τους καταναλωτές, για τους αγορές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις γενικά, πρέπει να είναι γενικότερα συγκρίσιμα αυτά τα επίπεδα. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση σχετικά διότι σε αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν καλύπτονται επακώς όλες αυτές οι πτυχές. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει αυτό, επειδή κάποιες κοινότητες και κάποιοι δήμοι έχουν ενδείξεις ότι κάποια οχήματα μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μπορούν να περνούν και να κυκλοφορούν στα αστικά κέντρα όταν πρόκειται για την διανομή κάποιων αγαθών, κάποιων εμπορευμάτων, για την ησυχία των καταναλωτών. Και στην Ολλανδία μόνο πολύ χαμηλής ηχοστάθμης ε, οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοια αστικά κέντρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η χορύπανση που προκαλείται. Γι' αυτό πρότασή μου labeling για τους καταναλωτές και τους αγοραστές. Σημαντικό στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, ένα πιο μακροπρόθεσμο χρονορίζοντα. Σε δύο βήματα περιορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την ηχορύπανση. Το τρίτο δεν είναι κλίμακα ουσιαστικά. Μετά από δύο και μετά από πέντε χρόνια προβλέπεται να γίνει κάτι. Αυτό όμω δεν είναι επαρκές και για τι εκπομπές ρήπων που είχαμε του διοξιδίου του άνθρακα είχαμε πρόταση διακομματικά ότι μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχοι πρέπει να ενταχθούν. Γι' αυτό και εδώ συνεκτικά εκφράζομαι υπέρ ενός πιο μακροπρόθεσμου στόχου για την μείωση της συγχωρήπανσης μακροπρόθεσμα σε ένα μεγαλύτερο χρονορίζοντα. Μετά από 14 χρόνια όλοι οι εμπλεκόμενοι έτσι μπορούν να ε, συντονιστούν και έγκαιρα να λάβουν υπόψη αυτά τα στοιχεία για το σχεδιασμό προϊόντων. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση. Η τρίτη πρόταση είναι μια διαφοροποίηση, περαιτέρω διαφοροποίηση των κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων και των οριακών τιμών έχει επικριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πολλές πλευρές και αναφέρθηκε αυτό πιο πριν. Και Σωστά αναφέρεται ότι οι κατηγορίες οχημάτων βασίζονται σε ένα παροχημένο ανεδαφικό σύστημα και γι' αυτό προτείνω σε σχέση με αυτό να έχουμε περαιτέρω κατηγορίες που θα ε, διεισδύσουν εδώ και όσον αφορά τι ε, τις ε, κατηγορίες 2, 3, N2, N3 να υπάρξει μια τέτοια διαφοροποίηση να ενταχθούν με διαφορετικό τρόπο με διαφοροποίηση αυτές οι ξεχωριστές κατηγορίες και σε διαφορετικούς τομείς γιοταχή και φορτηγά οι νέες κατηγορίες θα ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσει της τεχνολογίας και τις εξελίξεις της τεχνολογίας έχουμε λοιπόν την M3 σε τέσσερις κατηγορίες που διαφοροποιούνται επίσης και το N3 προτείνουμε δύο περαιτέρω κατηγορίες πέρα από αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίπτωση, οι οριακές τιμές μπορούν καλύτερα να προσαρμόζονται στην εκάστοτε κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων με ρεαλιστική προοπτική για τη μείωση της συγχωρήπανσης. Αυτό οδηγεί επίσης στο ότι κάποιες τιμές, οριακές τιμές, είναι πιο φιλόδοξου χαρακτήρα από ότι αυτές που εντάσσονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι στις διαφορετικές κατηγορίες, στο κατώτερο, στον κατώτερο τομέα διαφοροποιούμαστε πιο έντονα και πιο εξειδικευμένα. Και έτσι έχουμε ένα ρεαλιστικό επίπεδο ε, τιμών για την ηχοστάθμιση. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και διαμόρφωση των κατηγοριών, ώστε να έχουμε και καλύτερη διαμόρφωση και διαφοροποίηση των οριακών τιμών. Ένα στοιχείο θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Σε αυτό το νομοθετικό έργο πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλά νομοθετικά ως προτάσεις που αφορούν γιοταχή και φορτηγά οχήματα για αυτές τις διαφορετικές οδηγίες και κανονισμούς εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο και η μία επηρεάζει την άλλη. Έχουμε την Ευρω 5 και Ευρω 6, ε, έχουμε τον κανονισμό για τις εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα από τα ΙΟΤΑΧΗ και τα μικρά ε, φορτηγά ε, και έχουμε και απαιτήσει για την ασφάλεια. Πολλά όμως βρίσκονται σε αντίφαση το ένα με το άλλο. Τι συμβαίνει για παράδειγμα. Αν δεν έχουμε ένα νέο όχημα το οποίο να αναπτύσσεται από μηδενικό σημείο, διότι παίρνει πολλά χρόνια για να κλείσει ο κύκλος ζωής. Αν θέλουμε πιο πριν να μειώσουμε ε, κάποιες πτυχές, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όσον αφορά με παρέμβαση σε σχέση με τον κινητήρα. Αυτό τι γίνεται, τι κάνει. Κάνει, προσθέτει περισσότερο βάρος σε ένα τέτοιο όχημα, μηχανοκίνητο όχημα. Και τι γίνεται, σε ε, σαν μία πρώτη επίπτωση έχουμε μεγαλύτερη εκπομπή ρήπων. Όμω έχουμε πιο αυστηρέ διατάξει για τι εκπομπέ τρύπων. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε το ένα πράγμα επηρεάζει το άλλο και το ένα πράγμα να λαμβάνει υπόψη αυτέ τι ε, επιπτώσει που έχει σε άλλε πτυχέ. Για παράδειγμα, να μην δημιουργούμε προποθέσει που να δημιουργούν μεγαλύτερε εκπομπέ τρύπων που δεν επιτρέπονται. Αυτή την αλληλουχία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και μια άλλη πτυχή. Η σκάλα decibel αναπτύσσεται, εκτείνεται λογαριθμικά και όχι γραμμικά. Αυτό το έμαθα όταν ασχολήθηκα. 3 μείωση κατά 3 δεσιμπέλ ανταποκρίνεται σε 50% μείωση της ηχητικής επιβάρυνσης. Να το θυμόμαστε αυτό. Είναι λοιπόν μεγάλη η επίπτωση και η επιρροή, πράγμα το οποίο πάλι έχει επιπτώσεις στην τεχνολογία και στις τεχνικές προδιαγραφές. 6 δεσιμπέλ έχουμε 60% και με μεγαλύτερη ε, μείωση κατά 90% ε, ε, νέα προσαρμογή επιβάρυνση. Να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα για τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά οχήματα που θεωρούμε ότι είναι χαμηλών εκπομπών ρήπων. Έχουμε την πρόταση για την κατηγορία 1 να βρισκόμαστε πιο κάτω σε 67 δεσιμπέλ. Να τα θυμόμαστε όλα, όλα αυτά, να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές στις προσεγγίσεις μας, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό αποτέλεσμα. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, δύο σύντομες παρατηρήσεις για την έκθεσή μου ακόμα. Το πρώτο, έχουμε διαφορετικές φάσεις στην ανάπτυξη και σχεδιασμό όσον αφορά τα ΙΧ και τα φορτηγά. Γι' αυτό σε διαφοροποίηση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαφοροποιούμαστε και εμείς. Έχουμε 5 έως 7 χρόνια για τα ΙΧ, περίοδο σχεδιασμού, 8 και παραπάνω χρόνια για τα φορτηγά. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και το τελευταίο σημαντικό στοιχείο για την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή είναι το τεχνητό επίπεδο ε, θορύβων, τεχνικό ή τεχνητό επίπεδο θορύβων από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό το σημείο πρέπει να περάσει αφού εγκριθεί σε εμάς, από την πλευρά μας ε, να περάσει στην Ολομέλεια. Σε σχέση με τον κύριο Ούσκι υπήρξε υπόσχεση ότι θα συνεργαστούμε στενά. Η προσέγγιση μου είναι να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις που ίσως θα μπορούσαν να γελιοποιήσουν κάποιες προσεγγίσεις. Δηλαδή ποιο επίπεδο δεν θα έχει ένα ηλεκτρικό όχημα. Είναι αυτονόητα λοιπόν κάποια πράγματα. Ας μην υπερβάλλουμε. Έχουμε προσαρμόσει εδώ τους ορισμούς και αναφέρουμε ποιες ποια επίπεδα θορύβου μπορούν να είναι αποδεκτά. Ένα, ένας θόρυβος ε, όπως εκείνος που προκαλείται από ένα κινητήρα. Πρόκειται για εθελοντική υπόθεση, εθελούσια υπόθεση και ευθυγράμμιση. Όταν το κάνουν όμως αυτό και το λαμβάνουν υπόψη η παραγωγή, η, από πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, και να υπάρχει αντίστοιχη προσαρμογή για την ε, τροπολογία που έχουμε καταθέσει σε αυτή την κατεύθυνση στο ΧΕΒΗ. Και τώρα θα ήθελα ουσιαστικά να μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς να εισακουστεί η άποψή μας. Και ίσως και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα μπορούσε να δεχθεί τέτοιες προτάσεις. Ήδη συνεργαζόμαστε στενά. Αυτά για τα κυριότερα σημεία της έκθεσής μου. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές. Έχουμε και μια συνάντηση σκιωδών συντονιστών αύριο το απόγευμα και μπορούμε να δούμε αυτά τα θέματα του χρονοδιαγράμματος. Προσβλέπω συζητήσεις και τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα τους εισηγητές και καταρχήν την κυρία Βεστφάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν, η κυρία Βάισμπεργκερ αξίζει συγχαρητηρίων για την τοποθέτηση και τη γνωμοδότηση, διότι είχαμε πριν δύο εβδομάδες, αν δεν απατώμε, την πρώτη συζήτηση και νομίζω ότι οι στόχοι του σχεδίου της είναι σαφείς και απευθύνουν τα σωστά μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε ότι είχαμε συζητήσει στην πρώτη ε, φορά που ε, έγινε η παρουσίαση ή τι πρέπει να αλλάξει και ποια ε, σημεία κατακρίνουμε. Αλλά αυτό που είχα πει πριν δύο εβδομάδες έχουν περιληφθεί τώρα στην γνωμοδότηση πλην όμως ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να βελτιωθούν και εδώ σκέφτομαι ότι αύριο όταν θα μιλήσουμε για την ταξινόμηση, όταν μιλήσουμε για το εύρος που είναι αναγκαίο και την έκταση που είναι αναγκαία στο σημείο αυτό θα προβώ σε τροπολογίες εξού και τώρα θα σταματήσω εδώ διότι αύριο θα ε, ε, μπούμε στις λεπτομέρειες κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Άνια για την ευρία παρουσίασή της, διότι νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες συγκριωμένων συμφερόντων με άλλα θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και γι' αυτό μου αρέσει η προσέγγισή της. Καταρχήν ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το ε, υποβάλλει σαν κανονισμό. Εγώ είμαι υπέρ των κανονισμών και όχι τόσο υπέρ των οδηγιών διότι έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο μέλλον. Το, το, ο τομέας αυτός είναι πολύ καινοτόμος και πολύ σημαντικός για την Ευρώπη και νομίζω ότι έπρεπε να βελτιωθεί και να επιτύχει ένα διεθνές επίπεδο ε, ε, για να γίνει η Ευρώπη ένα είδος Silicon Valley που προωθεί ε, τα ηλεκτρονικά αλλά εμείς έχουμε ένα καινοτόμο τρόπο στην Ολλανδία που παρουσιάζουμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εις την Ευρώπη και ζητώ από την βιομηχανία να μας ενημερώσει ενημερώνουν ε, για τα, τις καινοτομίες τους που μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες. Ε, η Άνια είπε πολλά και έτσι δεν θα μακρηγορήσω. Το 1960 20% του πληθυσμού υπέφεραν από χορύπανση. Τώρα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ηλική, την ηχορύπανση και το επίπεδο που επηρεάζει το περιβάλλον, να συνδυάσουμε με άλλα είδη την αποδοχή των τύπων και είναι κάτι που πρέπει να συνδυάσουμε κατά τρόπον ώστε να μην ε, χρειάζεται να καταρτήσουμε νέα νομοθεσία. Και τέλος, αλλά δεν είναι το πιο επουσιώδες, είναι το σύστημα προειδοποίησεως του ΟΗΕ διότι στο ο Πεκίνο έχουν ε, προβλήματα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προκαλούν πολλά ατυχήματα γιατί ο κόσμος δεν τα ακούει να πλησιάζουν και είναι κρίμας. Γιατί αυτό που είπε η Άννα είναι ότι αποσύρω την ιδέα μου αυτή. Δηλαδή ε, ε, όπως βλέπετε ίσως θα έπρεπε να ακούμε τον ήχο των αλόγων που προχωρούν γιατί γιατί άλλαξε η νοοτροπία των ανθρώπων σχετικά με την αντιπετώπιση των μηχανών, των κινητήρων, αλλά χαιρετίζω και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, διότι όλοι θα συνεργαστούμε στα πλαίσια αυτά. Ευχαριστώ. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα ειδικό πάνελ όπου να κάνουμε τις ε, δοκιμές. Η κυρία Ρούλε, ε, σοβαρά, βρίσκω ότι η κυρία, Ρούλε, η κυρία ε, Βάισμπεργκερ πολύ σωστά παρουσιάζει τα θέματα, είναι της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, χαιρετίζω τις τροπολογίες της για την ενημέρωση των καταναλωτών καταναλωτών ε, και για τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτά που με προβληματίζουν και έχω υποβάλει γραπτές τροπολογίες είναι ότι ε, σε ορισμένους τομείς ξεπερνούμε την αρμοδιότητα της Επιτροπής και εδώ επιφυλάσσουμε διότι ε, θεωρώ ότι έχω πλέον κουραστεί από αυτές τις διαμάχες για την αρμοδιότητα των Επιτροπών αλλά την ευχαριστώ μέχρι στιγμής και για τις ιδέες και για την καλή συνεργασία.

Πρέπει εγώ τώρα να παρουσιάσω ορισμένα σχόλια σαν σκιώδης εισηγητή. Συμφωνώ με την γενική κατεύθυνση της προτάσεως, διότι όπως ξέρετε παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ στην εσωτερική νομοθεσία και πιστεύω ότι ένα βασικό θέμα για την πρόταση αυτή είναι ότι κινόμαστε ε, σε μεθόδους ε, δοκιμής του ε, θορύβου που θα ισχύσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει ε, να συγκρίνουμε τα ε, ε, τα αποτελέσματά μας με τα ισχύοντα ε, ε, πρέπει να καταλάβουμε γιατί έχουν επινοηθεί αυτές οι ε, δοκιμές διότι καλό είναι να υπάρχουν ορισμένοι θόρυβοι καλό είναι όμως να ρυθμίσουμε και το επίπεδο του θορύβου και του ήχου ε, επιπλέον, ε, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει παρουσιάσει αυτή η Επιτροπή είναι σχετικά με ε, τα τα οχήματα που έχουν χαμηλό επίπεδο θορύβου. Έχουμε ας πούμε τα οχήματα για τους αναπήρους, για, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες όπου υπάρχει μία χωριστή κατηγορία υποποίησεως και εδώ το πίσω μέρος των αυτοκινήτων το οποίο ε, πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε ράμπες ε, ε, επηρεάζει και τον τρόπο εκπομπών των καυσαερίων και θα πρέπει να συνδυάσουμε όλες αυτές τις ειδικέ τροποποιήσεις και κατά πόσον αυτά εκθέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Είναι λίγα ε, τέτοια οχήματα, χρησιμοποιούνται σε μικρές αποστάσεις, ε, δεν, ε, κάνουν, δεν χρησιμοποιούνται για πολύ μεγάλες κιλομετρικές αποστάσεις, οπότε πρέπει να εξετάσουμε και την αναλογικότητα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να υπάρξουν βελτιώσεις σε ορισμένους τύπους οχημάτων που δεν είναι αυτά που επιβαρύνουν περισσότερο την κυκλοφορία αντί αυτών που χρειάζονται να χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής. Πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των ε, κατασκευαστών ειδικών οχημάτων και εδώ υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε καταρτήσει ε, ειδικέ κατηγορίες για ορισμένα οχήματα και έχουμε δικαίωμα να τους ζητήσουμε να λάβουν υπόψη ότι αυτές οι εταιρείε δεν έχουν τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Προτού λοιπόν προχωρήσω θέλω να ρωτήσω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει την έκθεση της κυρίας Βάισμπεργκερ. Αν όχι, ε, ίσως... Ε, ζητήσω από την κυρία Μπονβιντσούτσο να απαντήσει και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαϊσγκιάδη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγήτες. Συνολικά γενικά μπορούμε να συμμεριστούμε τις προτάσεις σας και έτσι βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Για το θέμα προστασίας καταναλωτών και το labeling ήδη είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί, με ανοιχτό πνεύμα μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις. Η δική μας γραμμή και προσέγγιση είναι όπως ε, υπάρχει η δυνατότητα και για τα λάστιχα να ξεχωρίσουμε την έγκριση για τον τύπο και για το labeling. Το labeling όμως και τα στοιχεία πληροφόρησης ε, για τους καταναλωτές έχουν τη σημασία τους για τον τελευταίο στόχο, για τους στόχους θα πρέπει να υπάρχει συγκρισιμότητα και η σκοπιμότητα για την ανάλυση των στόχων για την βιομηχανία. Μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Να μην είναι επιζήμια για την προηγούμενη φάση την οποία υιοθετήσαμε και ταυτοποιήσαμε και διαρωτόμαστε για τον μακροπρόθεσμο στόχο το πρώτο βήμα θα ήταν για του νέου τύπου οχήματα και όχι για άλλες προσαρμογές ε, όπως και σε σχέση με προηγούμενες κατηγορίες. Για τις κατηγορίες οχημάτων ήδη το είπαμε. Είμαστε ανοιχτοί σε σχέση με προτάσεις ε, να δούμε αν υπάρχει ανάγκη πραγματικά να εξειδικεύσουμε κάποιες κατηγορίες ε, αυτοκινήτων ή οχημάτων σε σχέση με διαφορετικά, διαφορετικούς τύπους οχημάτων και να έχουμε έναν πιο σωστά επιμερισμένο ε, στόχο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρότασή σας, να δούμε δικαιολογείται ή όχι αυτή η εξειδίκευση ή σε σχέση με πολλές κατηγορίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Κατανοούμε όμως την λογική του να έχουμε εξειδίκευση όσον αφορά και τα εμπορικού χαρακτήρα οχήματα. Θα αναφέραμε ιδιαίτερα εκείνα τα οποία θα ήταν για τη μεταφορά επιβατών για παράδειγμα και όχι τόσο για μεταφορά αγαθών. Για τις ε, επιχειρήσεις ε, είμαστε ευαίσθητοι για αυτό το θέμα που έχει ήδη συζητηθεί. Είναι ένα από τα θέματα όπου υπάρχει συμφωνία σε σχέση με την ομάδα εργασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διαφοροποιήσεις και να δούμε σε σχέση με τις διαφορετικές διατάξεις, νομοθετικές διατάξεις, να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Μπορούμε να εξετάσουμε και να δούμε αν είναι σκόπιμο για την ανάλυση κόστους-οφέλους να έχουμε διαφορετική και τέτοιες διατάξεις ε, για τη μεταφορά επιβατών, για, την, για τα οχήματα μεταφοράς αγαθών, ανάλογα με τις ε, εξειδικεύσεις. Προσπαθήσαμε για αυτή την εξειδίκευση να ευθυγραμμιστούμε περισσότερο με την ε, υφιστάμενη ρύθμιση. Έχουμε συμπεριλάβει και μία δυνατότητα υπό την πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται αυτό και για τα ηλεκτρικά οχήματα υπό τις διατάξεις για την, ηχητική, για την παραγωγή ε, ήχων από αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα με βάση αυτά που συμφωνήθηκαν και εκπονήθηκαν στη Γενέβη. Θα υπάρχει ενημέρωση και επικαιροποίηση αυτών ώστε να λαμβάνουμε υπόψη κάποιες τεχνικές εξελίξεις ή οποιασδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις που συμφωνούνται στην Γενέβη για τον χαμηλό όγκο ιδιαίτερα εκείνων των οχημάτων που θεωρούμε υπό την οδηγία πλαίσιο, μια και έχουμε εδώ και την έγκριση τυπολογίας ή τύπων, πρέπει να επικαιροποιούνται οι διατάξεις ε, για τέτοιου είδους μικρά οχήματα και για τα αστικά κέντρα και μια μείζον επικαιροποίηση όσον αφορά αυτά είναι εκείνη που βρίσκεται υπό εξέλιξη και που σύντομα θα καλυφθεί με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα τον λόγο στην κυρία Βάσκερμπορ για να μας συνοψίσει και για να μας επιβεβαιώσει και το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Βάσκερμπορ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδει εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ιδιαίτερα επικοδομητικό πνεύμα. Θέλω να συνοψίσω ω εξή το ότι το βρίσκω ικανοποιητικό. Τουλάχιστον αυτές είναι αυτά τα πρώτα μηνύματα. Και υπάρχουν κάποια σημεία που με κοινέ τροπολογίε μπορούν να καλυφθούν ή υπάρχει και η προθυμία από πλευράς μας να τα ρυθμίσουμε έτσι και για το labeling. Ειδικά πιο πριν είπα ότι δεν το έχω εντάξει στο χαρτοφυλάκιο αυτό, διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ξεχωρίσουμε αυτά τα θέματα και νομοθετικά, αλλά υπάρχει η πρόθεση και επιθυμούμε κι εμείς να υποβάλει μια τέτοια πρόταση για το labeling η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκόπιμο θα ήταν αυτό το labeling να λαμβάνει υπόψη και τα labeling για την ετικετοποίηση ή τις ρυθμίσεις για την εκπομπή ρήπων. Να μην έχουμε ξεχωριστά στοιχεία κάθε φορά για τις εκπομπές ρήπων, για την ηχορύπανση. Να μπορούν όλα αυτά να εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο και να υπάρχει συνεκτικότητα και συνάφεια. Είναι θέμα προστασίας καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάσσεται. Για τα ηλεκτρικά οχήματα δεύτερο. Έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι για την, τον ορισμό της Γενέβης ε, που χρησιμοποιήθηκε το βρήκα όμως κάπως ατυχές τόσο εξειδικευμένα ή μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να περιοριζόμαστε Ίσως μπορούμε και με μια άλλη διατύπωση να ε, προχωρήσουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα σε λεπτομέρειες, ε, σε διαφορετικές πτυχές. Ήταν σημαντικό όμως να προταθεί μια προτα... ένας ορισμός όπου να απόσχουμε από αυτή την εξειδίκευση, την υπερβολική εξειδίκευση. Διότι κάποιοι συνάδελφοι, για παράδειγμα, θα προτιμούν κάποιες, ε, κάποιοι ήχοι από ζώα, όπως προαναφέρθηκε από τον συνάδελφο Μάντες, να μην εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Μπορούμε όμως νομίζω να συμφωνήσουμε για τις κατηγορίες, κατηγορίες οχημάτων, για τη διαφοροποίηση τώρα, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε κατανοητό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, μεγαλύτερη προσαρμογή στις, ε, στα χαρακτηριστικά των επιμέρους αυτών προϊόντων. Έχω ανοιχτό πνεύμα να δούμε αν το ένα ή άλλο μπορεί να εξαιρεθεί ή να συμπεριληφθεί ώστε να υπάρχει απλούστευση και λειτουργικότητα. Είναι σημαντικό όμως να προσαρμοζόμαστε στο τρέχον, στην τρέχουσα φάση της τεχνολογίας επικαιροποιημένα. Και συνάδελφε Χάρμπορ, είμαι πρόθυμη το θέμα των ειδικών οχημάτων να το εξετάσουμε και όλες τις άλλες παρατηρήσεις που έγινε, έγιναν. Να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Ήταν σημαντικό για μένα να δούμε ποια είναι τα οχήματα εκείνα που από πλευρά όγκου δημιουργούν κάποιε ξεχωριστέ καταστάσει και να δούμε τι ε, οριακέ τιμέ και να δούμε αν επαρκεί μια κατηγορία ή η άλλη. Διότι έχουμε και κάποια επίπεδα τα οποία είναι πιο αυστηρά ίσω σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι πρόθυμη να τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ για την καλή θετική ανταλλαγή απόψεων. Να επισήσω την προσοχή σα στο χρονοδιάγραμμα. Αύριο, την Τετάρτη, από τι 2 στι 3 το μεσημέρι, το απόγευμα, θα έχουμε συνάντηση οδόν εισηγητών. Μετά θα έχουμε την προθεσμία, καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι και στις 20 ε, Ιουνίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Στις 21 Ιουνίου έγκαιρα θα ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία, στην, θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στις 21 Ιουνίου θα πρέπει να έχουμε την ψηφοφορία εμείς εδώ να μην γίνει η ψηφοφορία δηλαδή μια μέρα πριν από εμά, να έχουμε χρόνο με την ψηφοφορία να λάβουμε υπόψη αυτή την έκθεση. Και είμαι και μέλο στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και αυτέ τι σκέψει θα τι εκθέσω και στην ίδια την Επιτροπή Περιβάλλοντο να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή Κομισιόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ας προχωρήσουμε στα δύο τελευταία θέματα τη σημερινή διάταξη που θα τα εξετάσουμε μαζί. Υπάρχει χρόνο μέχρι τις 12.30 για να συζητήσουμε αυτές τις πολύ σημαντικές εκθέσεις για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Ο φίλος και συνάδελφος Λουί Κρέκ δυστυχώς είναι στο νοσοκομείο και τώρα αναρρώνει σπίτι του. Και αυτό είμαι βέβαιος ότι εξ τη Επιτροπής μπορούμε να το ευχηθούμε περαστικά Ευχαριστώ πολύ. Και part, Wellpart ε, λάβει τη θέση του και κατόπιν έχουμε ε, την κυρία Σουν, ε, την εισηγήτρια, που θα μιλήσει για το δικό της θέμα και μετά τους σκιώδεις εισηγητές για τις διάφορες εκθέσεις. Λοιπόν, όταν, ή μάλλον, αυτό το οποίο προτείνω να κάνουμε είναι το εξής, με την αδειά σας. Θα καλέσω τους δύο εισηγητές να μας κάνουν τις παρουσιάσεις τους και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια και για τις δύο εισηγήσει. Ο κύριος δεν είναι εδώ. κύριος Κύριο Ρέκο. κύριος Ροσφόρ και για τις δύο εκθέσεις. Κύριε Ρούλη και τις δύο. Κύριος Πόψη και για τις δύο. Ο κύριος Διόμ δεν είναι εδώ, νομίζω. Λοιπόν, με χαρά καλωσορίζω τον Χριστίνα Γιούτο, την επικεφαλής μονάδος που ήταν πάρα πολύ δραστήρια και γνωρίζω ότι έχει δει όλου του συγητέ. γι' αυτό θα της δώσω ε, το λόγο μετά από τον πρώτο γύρο των συζητήσεων. Έχουμε δύο σχέδια εκθέσεων τα οποία θα έχουμε υπόψη και καλωσορίζω επίσης και την Προεδρία της Δανίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αλφαβητική σειρά, με το ADR πρώτα, την κυρία Γκέπαρτ, να παρουσιάσει ε, την έκθεση του κύριου Γκρέπτ εξ ονόματός του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την Παρασκευή τηλεφώνησα με τον κύριο Γκρέκ και είναι και ανυπόμονος και θέλει να επιστρέψει με κάθε τρόπο, ξέρετε, τη δουλειά αυτή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οι γιατροί όμως του σύστησαν να παραμείνει στο σπίτι του και θέλει όμως να επανέλθει και γι' αυτό θα είμαι εγώ τώρα η εισηγήτρια εξ ονόματός του. Μου έστειλε τις σημειώσεις του και έτσι μπορώ να το κάνω αυτό. Ξεκινά με το περιεχόμενο της έκθεσης και τα πλαίσια στα οποία βρίσκεται αυτό, αυτή η ουσία. Είναι για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικό να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκούν τα δικαιώματά τους με ελεύθερο τρόπο, χωρίς περιορισμούς. Και σε αυτό ανήκει φυσικά η δυνατότητα να μπορούν να έχουν προϊόντα και υπηρεσίες στη διάθεσή τους που θα μπορούν να αγοράζουν στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της χώρας τους έμεσα ή άμεσα και μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, του δικτύου, ηλεκτρονικού δικτύου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες αυτές οι πτυχές σε αυτό το θεματικό φάσμα, θεματολογικό φάσμα. Φυσικά οι δυνατότητες αυτής της ελευθερίας στα κράτη-μέλη όσον αφορά προσπελασιμότητα η ποιότητα, πολλές φορές υπάρχουν κενά και προβλήματα και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις πρώτες συστάσεις της ήδη πριν από 14 χρόνια για την την προσέγγιση αυτών των θεμάτων για τους καταναλωτές και την ρύθμισή τους. Όμως η υλοποίηση ή τα μέτρα τα οποία έλαβαν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο είναι εμβαλωματικά, είναι ένα patchwork μεταξύ ADRs και δεν συντεριάζουν όσον αφορά και το ποιοτικό επίπεδο και την ε, προσπελασιμότητα, την ε, δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά οι πολίτες και είναι πολύ διαφορετικού χαρακτήρα εκάστοτε. Γι' αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προχωρήσουμε και ευρωπαϊκά να ρυθμίζονται αυτά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη μελέτη επιπτώσεων προχώρησε σε, σημαντική, σε ρύθμιση σημαντικών θεμάτων που την χάνουν απαντήσεων τώρα και που πρέπει να ρυθμιστούν ευρωπαϊκά. Μεταξύ αυτών είναι, συγγνώμη, το κείμενο είναι στα αγγλικά. Τα αγγλικά μου όμω δεν είναι τόσο καλά και γι' αυτό δεν μπορώ να τα εκφράσω αγγλικά. Γι' αυτό μεταφράζω ε, από τα αγγλικά στα γερμανικά. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια προβλήματα στι εκφράσει μου. Υπάρχουν τα εξή που πρέπει να βρούμε λύσεις. Η κάλυψη τομεακά και γεωγραφικά κάποιων τομέων. Η, πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες για τα ADRs και η διαφορετική ποιότητα για την δυνατότητα επιδιαιτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Η επιδιαιτησία, η αντιμετώπιση δηλαδή τριβών και προβλημάτων, τι σημαίνει οι Ευρωπαίοι, οι καταναλωτές μόνο τότε θα μπορούν διασυνοριακά να αγοράζουν τέτοια προϊόντα όταν θα είναι αξιόπιστα αυτά, σε αξιόπιστα πλαίσια. Και αν είναι αναγκαία και χρειαστεί να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες τριβές και προβλήματα με μια επιδιαιτησία ή ας το πω έτσι εξοδικαστική ρύθμιση προβλημάτων. Είναι σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν πολλούν διασυνοριακά επειδή πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τι θα γίνει αν υπάρχει θέμα τριβών και προβλημάτων. Πώς θα ε, ε, ρυθμίζονται ε, και ποια επιδιαιτησία θα υπάρχει για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων δεδομένου του διαφορετικού πλαισίου κάθε φορά που ισχύει από κράτος σε κράτος και για το online banking και για το online αγορές ηλεκτρονικές και ε, συναλλαγές ε, τραπεζικές που θα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε όπως θα έπρεπε όλες αυτές τις δυνατότητες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο παράλληλα με την ε, επιδιατησία να υπάρχει και μια ODR πλατφόρμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά. Και το ODR και το ADR είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό και τα δύο αυτά παράλληλα να ρυθμίζονται. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή πρωτοβουλία, μια καλή πρόταση. Χρειάζεται όμως ακόμα κάποιες βελτιώσεις ε, που πρέπει να προβλεφθούν για να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των συστημάτων και των πλαισίων αυτών και των ε, οργάνων και όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους και το αξιόπιστο του έργου τους και να είναι λειτουργικές αυτές οι δράσεις διαφανείς και αποτελεσματικές. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε για το πεδίο εφαρμογών. Και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι καταναλωτές είναι οι καταναλωτές που έχουν κατοικούν και έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια αμερόληπτη, ουδέτερη όσον αφορά την ε, επίδρασή της ε, υπηρεσία επιδιαιτησίας και ρύθμισης που πρέπει να είναι αποτελεσματική διασυνοριακά cross-border και το ίδιο το κράτος μέλος ε, στο οποίο ασκείται μια τέτοια ε, προσφυγή ή μια τέτοια, αναλαμβάνεται μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να μπορούν να δράσουν. Για αυτή την οδηγία, ευχαριστώ κύριε Σβάπ που με βοηθήσατε με τον όρο, οδηγία έψαχνα να βρω. Αυτή η οδηγία πρέπει και αυτές τις δύο ανάγκες να καλύπτει. Διασυνοριακά και εθνικά, εθνικές ε, περιπτώσεις. Διασυνοριακές και εθνικές. Αυτό έχει τεράστια σημασία πρέπει εκ παραλίλου να δράσουμε. Τώρα, μία δράση ή μία αποκλειστική εφαρμογή διακρατική ή διασυνοριακή, δηλαδή διαφοροποίηση εθνικών υποθέσεων και διασυνοριακών δεν θα ήταν θετική υπόθεση. Γιατί αν είχαμε ξεχωριστές ρυθμίσεις θα είχαμε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό των ADR και θα είχαμε άνισο επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκρέκ θα συνιστούσε να μην κάναμε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Γκρέκ στην έκθεσή του προτείνει και κάτι άλλο. Μας προτείνει η καταναλωτές ε, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ε, σε αυτές τις ε, ε, δυνατότητες, όχι οι επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις έχουν και άλλες δυνατότητες και άλλα μέσα στη διάθεσή τους. Θα είναι καλό λοιπόν να αποσαφηνίσουμε και να πούμε ότι μόνο για πολίτες καταναλωτές θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα των ADRs. Να μην υπερφορτώσουμε δηλαδή και με τις επιχειρήσεις ε, αυτές τις ε, υπηρεσίες. Τώρα όσον αφορά την πρόσβαση προς πελασιμότητα στις ADRs θα πρέπει να είναι στην πρόσβαση προσπερασιμότητα όλων των καταναλωτών που κατοικοεδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό προτείνεται σε αυτή την έκθεση τα κράτη-μέλη την πρόσβαση αυτή να την ρυθμίζουν και την ποιότητα των ε, υπηρεσιών αυτών να την αναβαθμίσουν, να διασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας καταναλωτών με αυτές τις βελτιώσεις. Επιπλέον πρέπει να προβλέψουμε επιπρόσθετα εύκολη προσπελασιμότητα σε πληροφορίες και στη διάθεση πληροφοριών και στην δυνατότητα όταν ζητηθεί να υπάρξει παρέμβαση επιδιαιτησίας. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες να βελτιωθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικά μεγάλο εύρος άρνησης ε, επιδιατησίας για να μην ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα και υπάρχει δυνατότητα μετά να παρακάμπτονται οι διαδικασίες αυτές, οι διεργασίες επιδιατησίας. Σημαντική υπόθεση για τον κύριο Γκρέκ αυτό. Επιπλέον έχει και μια τροπολογία που έχει προετοιμάσει και καταθέσει ο κύριος Γκρέκ, όπου το αποτέλεσμά της θα ήταν αν και όταν ένας καταναλωτής θέλει να κάνει χρήση δυνατότητας επιδιατησίας αυτό δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα του προσφυγή σε αστικά δικαστήρια, διότι μπορεί να προβλέπονται κάποιες διαδικασίες ή χρονοδιορίες, ε, ας το πω έτσι, προθεσμίες που δεν πρέπει να περιορίζουν τέτοια δικαιώματα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανεξαρτησία αυτών των υπηρεσιών και φορέων και ο κύριος Γκρέκ έχει προετοιμάσει και καταθέσει μια τροπολογία που παράλληλα με την αμεροληψία και την ουδετερότητα προβλέπει και τονίζει την ανεξαρτησία των αρχών επιδιαιτησίας ώστε πραγματικά να υπάρχει σκοπιμότητα στην χρήση, αποτελεσματικότητα στην χρήση αυτών των υπηρεσιών και να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στις υπηρεσίες που παρέχουν οι δυνατότητες επιδιαιτησίας. Πρέπει να είναι βέβαιοι οι καταναλωτές, να υπάρχει ασφάλεια, νομική ασφάλεια για αυτούς ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτές τις ε, υπηρεσίες. Ένα άλλο θέμα είναι η διαφάνεια. Υψηλότατος βαθμός διαφάνειας πρέπει να διασφαλίζεται. Όχι μόνο την αξιοπιστία θα την βελτιώνει η αυξημένη διαφάνεια και για τους ε, εμπόρους και για τους καταναλωτές, αλλά επίσης και οι αναγκαίες πληροφορίες θα διαχέονται και τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα διαφανές πλαίσιο που θα οδηγεί σε ένα σωστό πεδίο εφαρμογής των δυνατοτήτων επιδιαιτησίας. Επιπλέον αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Αυτές οι υπηρεσίες και οι φορείς τους πρέπει να είναι αποτελεσματικές, απλές, να μπορούν γοργά να δράσουν και να μην επιβαρύνουν με ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Είναι τρία κριτήρια που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο Γκρέκ. Τα EDS θα πρέπει την επιδιαιτησία να την διασφαλίζουν σε περίοδο τριών μηνών το πολύ, εκτός αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα περίπλοκα και τεχνικά ιδιαίτερα δαπανηρά θέματα που θα απαιτούν ε, ειδικέ διεργασίες. Να μην, περνάμε να μην ξεπερνάμε την προθεσμία των τριών μηνών, 90 ημερών για να είμαστε αποτελεσματικοί. Για να καταστούν όλα αυτά εφικτά, πρέπει γοργά να μπορούν οι καταναλωτέ να έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε ADR. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει χωρίς τέλη και επιβαρύνσεις να γίνεται αυτό. Αν υπάρχουν κάποια τέλη όμως και επιβαρύνσεις, ε, ε, οι εισφορές θα πρέπει να είναι σε ένα λογικό πλαίσιο που δεν θα δημιουργούν, ας το πω έτσι, υπερβολική επιβάρυνση για τους πολίτες. Μετά, νομική ασφάλεια και βεβαιότητα για τους καταναλωτές. Ο κύριος Γκρέκ εδώ τι λέει. Εισάγει την αρχή της ελευθερίας, συμβατικής ελευθερίας για τους συμβαλόμενους. Αυτό πρέπει να το εννοήσει κανείς ως εξή. Ακόμα και όταν υπάρχει επιδιαιτησία, ακόμα και όταν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα επιδιαιτησίας, παρόλα αυτά πρέπει να είναι ελεύθερος ένας καταναλωτής αν τον δυσαρεστεί αυτή η, το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας επιδιαιτητικής ε, διασφάλισης των συμφερόντων του πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει στα δικαστήρια αν το επιλέγει, ώστε η νομική ασφάλεια ασφάλεια και η νομική βεβαιότητα να κατοχυρώνεται, ιδιαίτερα στους διασυνοριακούς τομείς και συναλλαγές, εκεί όπου οι καταναλωτές για την νομική ασφάλεια δεν θα πρέπει να αποκλείονται όσον αφορά νομική ασφάλεια που δημιουργείται από το εθνικό σύστημα των εθνικών κρατών μελών. Αυτές οι δύο αρχές διασυνοριακών συναλλαγών και εθνικής βεβαιότητας ε, νομολογίας πρέπει να ε, βαίνουν εκ παραλίλου. Αμφότερες οι πλευρές πρέπει να είναι θετικά καλά ενημερωμένες και να μπορούν έτσι να αποφασίζουν αν θα δέχονται μια τέτοια ένα δεσμευτικό πλαίσιο ε, απόφασης και νομολογίας. Αν δεν το δέχονται θα πρέπει να απορρέει η ε, συμβατική ελευθερία, η ελευθερία των συμβαλωμένων να επιλέγουν προσφυγή σε αστικά δικαστήρια. Προτού δηλαδή καταστεί αναγκαία μια τέτοια επιδιαιτησία για ένα οποιοδήποτε θέμα, ο καταναλωτής πρέπει ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα μιας τέτοιας επιδιαιτησίας να μπορεί να το αποδεχτεί, αλλά δεν είναι αποκλειστικά δεσμευτικό κάτι τέτοιο εκ προημίου μπορεί στο τέλος να αποφασίσει λόγω της ε, ε, ελευθερίας, της συμβατικής ελευθερίας που θα διασφαλίζεται να ασκήσει περαιτέρω δικαιώματα για την ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων του αυτών παράδειγμα νομική τέτοια προσφυγή αν δεν ικανοποιείται για τα θέματα πληροφοριών, πληροφόρησης συμβαίνει το εξής πολύ λίγοι πολίτες γνωρίζουν για τα υφιστάμενα μέσα και αρχές επιδιαιτησίας μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική υπόθεση να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να μεριμνήσουμε να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες να πληροφορούνται σωστά το τι συμβαίνει και τι τους προσφέρεται. Γι' αυτό το άρθρο 10 έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου απαιτείται μέσω του άρθρου αυτού ή καταναλωτές από τους ίδιους τους εμπόρους να ενημερώνονται ότι υπάρχουν τέτοια κομβικά σημεία ε, για την επιδιαιτησία. Να μην παραμένουν δηλαδή, να μην υπάρχει άγνοια πλέον, αλλά να ενημερώνονται. Και αυτή η απέτηση της πληροφόρησης και ενημέρωσης από τους ε, εμπόρους ε, και επιχειρηματίες δεν πρέπει να είναι γραφειοκρατικά δίσκαμπτη ώστε να πιέζονται οι καταναλωτές εδώ λοιπόν σε εξειδικευμένες προτάσεις που υποβάλλονται προβλέπεται η ρύθμιση αυτή ώστε να διευκολύνει τους καταναλωτές. Ζητείτε επίσης παρακαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές ως προς ανατολισμούς ώστε να να υπάρχει αποσαφήνιση και βελτίωση για την λειτουργία αυτής της οδηγίας και βελτίωση της νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας. Και ζητεί να υπάρξει και monitoring, εποπτεία, επιτήρηση για όλες αυτές τις διεργασίες, για την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή και ε, συμμόρφωση με τις αρχές αυτής της οδηγίας, πράγμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί σωστά. Ολοκληρώνοντας, υπάρχει, έχει ο Λουί Γκρέκ εδώ ένα, σε τρεις άξονες, σε τρεις πυλώνες, ε, μια σε τρεις πυλώνες πρόταση η ε, τα κενά που υπάρχουν μέσω των ADR πρέπει να ξεπεραστούν να καλυφθούν σωστά, ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο που θα δημιουργηθεί για τους καταναλωτές. Να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές σε όλους τους τομείς τομεακά και γεωγραφικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση διατομεακά σε δυνατότητες επιδιαιτησίας. Να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα. Η υπέρβαση των κενών, των ελλείψεων όσον αφορά πληροφορίες και άλλα προβλήματα έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Και τέλος ο εναρμονισμός. Ο εναρμονισμός όσον αφορά το κριτήριο της ποιότητας, της αναβάθμισης ποιοτικά αυτών των θεμάτων από τους αρμόδιους για την επιδιαιτησία. Η επιδιαιτησία πρέπει να έχει υψηλή ποιότητα, να είναι αναβαθμισμένη, να είναι αμερόληπτη, διαφανής και αποτελεσματική. Έχουν τεράστια σημασία αυτά. Υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία ίσως είναι επίμαχα στην ε, εξέτασή τους. Το άρθρο 2α για παράδειγμα, α, 2αα, τι γίνεται εδώ για το πεδίο εφαρμογής, το εύρος εφαρμογής αν τα άτομα, για παράδειγμα, τα οποία είναι αρμόδια για τα θέματα ADR, αν θα ε, την χάνουν μισθού, αν θα πληρώνονται γι' αυτό ή όχι. Το άρθρο 8 για την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα. Ο Λουί Γκρέκ τι προβλέπει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 90 ημέρες προθεσμία να προβλέπει κατά το μέγιστο ως χρονικό όριο για την ρύθμιση τέτοιων τριβών και προβλημάτων. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε μήπως μπορεί να ρυθμιστεί σε μικρότερη χρονική περίοδο, μικρότερη των 90 ημερών. Το άρθρο 10, πληροφόρηση ενημέρωση πώς όλα αυτά τα θέματα θα παρέχονται ως πληροφορίες, ως στοιχεία στους καταναλωτές. Ο κύριος Γκρέκ τι προτείνει εδώ. Προτείνει να μην είναι υποχρεωτικά σε κάθε λογαριασμό να αναφέρεται αυτό, αλλά στις προσυμβατικές διατάξεις πριν από το τελικό συμβόλαιο ή σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο αλλά να είναι προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες και να υπάρχει ένα περιθώριο στους εμπόρους πώς θα διανέμουν, πώς θα διαχέουν αυτές τις πληροφορίες προς τους πελάτες, τους καταναλωτές. Να μην υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση. Δεν θέλουμε ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν προβλήματα λόγω γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και προσκομμάτων και εμποδίων γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Και τέλος, τα κράτη-μέλη, τέλος, τέλος, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τα ίδια να συζητήσουν και να ρυθμίσουν να δουν πώς αυτό το πλαίσιο επιδιαιτησίας θα ακολουθεί ειδικού κανόνες, ξεχωριστές διεργασίες, ώστε να καλύπτονται οι πτυχές αποτελεσματικά. Ελπίζω ότι τα απέδωσα σωστά αυτά τα οποία σημείωσε ο κύριος Γκρέκ και ήθελε να σας τα εκθέσω. Προσβλέπω να ακούσω τις απόψεις και αυτά τα οποία θα πει και η κυρία Τούν και θα τα διαβιβάσω όλα στον κύριο Γκρέκα. Ευχαριστώ. thank you very much. Ευχαριστώ. Και πάλι ε, παρακαλώ διαβιβάστε τις ε, ε, ε, ε, ε, όλες μας τις ευχές στον κύριο Γκρέκ. Σημειώσαμε αυτά που πρότεινε και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Τέν η οποία θα παρουσιάσει τη δική της έκθεση και μετά θα σας παρακαλούσα να τελειώσουμε στις 12 γιατί χρειάζονται οι σκιώδεις κάποιο χρόνο να παρουσιάσουν αλλά η κυρία Τέν ας παρουσιάσει την πρόταση έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ήταν ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία και με τον Λουί Γκρέκ ε, ε, συναντηθήκαμε επανειλημμένως διότι θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ρουσό που είναι εδώ σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε για τα ADR και ODR. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφοροι εδώ οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα αυτό και που αποδεικνύει ε, ότι ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να ε, συμβάλλει σε την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν και οι πολιτές και οι καταναλωτές είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον τρόπο εμπορικών συναλλαγών διότι μόνο, ιδίως διασυνοριακά όπου μόνο 9% των Ευρωπαίων αγοράζουν διασυνοριακά 12% θεωρούν ότι είναι ασφαλείς όταν αγοράζουν διασυνοριακά και οι υπόλοιποι λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κατήρτισε ε, μία νομοθετική πρόταση κατά τρόπον ώστε να βελτιώσει την κατάσταση και εγώ έτσι την αξιολογώ και με αυτό το πνεύμα την πρόθυσα. Θέλουμε δηλαδή να βελτιώσουμε την κατάσταση και ιδίω να ξαναδώσουμε ε, στους πολίτες και καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εμπιστοσύνη στην αγορά. Ε, να υπάρχουν δηλαδή περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές γιατί θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου. Η πρόταση έχει υποβληθεί και η στάση μου επ' αυτής είναι ότι συμφωνώ με τον κύριο Γκρέχ, δηλαδή τα ADR πρέπει να είναι σαφή. Αλλά αυτή η πλατφόρμα ODR, δηλαδή εξοδικαστική επίλυση των διαφορών, ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχουν καν ακούσει οι καταναλωτές, δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και οι πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτών των ρυθμίσεων. Δεν χρειαζόμαστε ένα άλλο, μια άλλη πύλη ηλεκτρονική για πληροφόρηση, αλλά να την εντάξουμε σε μια ισχύουσα και υπάρχουσα πύλη ηλεκτρονική. Αυτή ήταν η αντίδραση που εγώ εισέπραξα. Θα πρέπει να περιληφθεί στην πύλη Europe, η οποία υπάρχει ήδη, να υπάρχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση για όλους τους πολίτες που θα μπορούν και να πληροφορηθούν και να βοηθηθούν. Επίσης ε, νομίζω ότι δεν πρέπει απλώς να διευρύνουμε το, την εμβέλεια αλλά ε, το, να μπορεί η ρύθμιση αυτή ODR να ισχύσει όχι μόνο ε, διασυνοριακά αλλά και ενδοσυνοριακά και να αποφασίζει ο καταναλωτής τι θέλει να επιλέξει να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επανόρθωσης εάν ο καταναλωτής δεν βρει μία λύση με τον πολιτή. Πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ε, μεγαλύτερα τμήματα στην ενιαία αγορά εφόσον δεν έχουμε σύνορα στην ενιαία αγορά μεταξύ των κρατών και πρέπει να υποχρεώσουμε ε, τους εμπόρους να λάβουν υπόψη τις ρυθμίσεις αυτές, να ε, προωθούν ε, μία διασύνδεση προς μία ηλεκτρονική διεύθυνση με μία πληροφορία ή με ένα κουμπί που μπορεί εύκολα να βρει ο καταναλωτής και θα του διοχετεύει δημοσιεύεται και από τον έμπορο. Αυτό που ονομάζουμε διεύρυνση της εμβελίας, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε διαφορετικά, αλλά η διεύρυνση της εμβέλειας σημαίνει ε, σχετικά με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, είναι ε, η δυνατότητα να δώσουμε ε, μία διεύθυνση ή στον καταναλωτή που θα μπορεί να επιλύει όλες τις διαφορές και θα έχει πολλά προσόντα σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της ενιαίας αγοράς και θα συνεπάγεται ελάχιστο ε, επιπρέωστε τη χρέωση ιδίως για αυτούς που χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα για διάφορες περιπτώσεις Οπότε ε, θα μπορεί κανείς ε, ε, έτσι με το ίδιο κόστος να καλύψει και τις ενδοσυνοριακές και εσωτερικές διαφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της έχει διατυπώσει ορισμένες πληροφορίες ε, για το πόσο θα πρέπει να αντιδρά ο ενάγων ε, και πρέπει να δω το πρότυπο αυτής, ε, αυτού του εντύπου. Θέλω δηλαδή να δω πώς θα προχωρήσουμε και πόσα αυτοί οι οποίοι παραπονούνται ε, μπορούν ε, να ε, παράσχουν πληροφορίες, τι επαφές πρέπει να υπάρξουν μεταξύ της πλατφόρμας διαχειρήσεως των παραπώνων με τον καταναλωτή και νομίζω ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να επιζητήσει τέτοιες λύσεις. Επίσης τα ODR βασίζονται σε μία μεταφραστική μηχανή την οποία δεν έχουμε δει ακόμη. Είναι αυτόματη μετάφραση που είναι πολύ σημαντικό θέμα που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ε, πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ζητούμε μία κατεξουσιοδότηση πράξη για να δούμε πόσο θα λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα για τις προθεσμίες. Νομίζω ότι 90 ημέρες είναι πάρα πολύ μακρύς χρόνος, αλλά επειδή οι τρόποι αυτοί επιλύσεων των διαφορών ADR και ODR θα πρέπει να συμβαδίζουν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και ε, προτείνουμε ε, για τη διαδικασία ODR ένα χρονικό περιθώριο 7 εργασίμων ημερών και για όλη την ε, διαδικασία θα πρέπει να καλύπτεται σε 90 μέρες όπως είναι τα ADR που μου φαίνεται μακρύ αλλά σε πολλές χώρες κρατά πολύ περισσότερο και μια δικαστική επίλυση των διαφορών θα διαρκούσε επί χρόνια χρόνια. Γι' αυτό και έχω προσπαθήσει να προβώ σε πιο ουσιαστικές αλλαγές, όχι μόνο διασυνοριακά, αλλά να υπάρχει και ένα σύστημα πληροφόρησης εσωτερικό, εθνικό και έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες μέχρι τέλη Μαΐου και η πληροφόρηση αυτή νομίζω ότι και από πλευρά του κυρίου Γκρέχ εφόσον έχουμε συνεργασία επί του θέματος είναι πολύ ουσιαστική και η γλώσσα είναι επίσης βασική δεν είναι μόνο η χώρα ε, όπου είναι εγκατεστημένος ο καταναλωτής αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιεί δεν σημαίνει ότι επειδή ζει σε μια χώρα χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα και δεν είναι υποχρεωτικό η γλώσσα να είναι αυτή του χώρου διαμονής της χώρας διαμονής. Και επίσης όπως σας είπα θα πρέπει να υπάρχει ένα έντυπο εγώ προτιμώ να μιλάμε ε, για ε, συμβούλους ε, για την επίλυση διαφορών και τέλος προτιμώ τα ODR να καλύπτονται από το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών που θα μπορούν να περιλάβουν και τα εθνικά σημεία επαφής για ODR, οπότε θα είναι ακόμη πιο πλήρης η ενημέρωση. Και θέλω να προσθέσω μία πληροφορία. Μιλάμε τόσο πολύ για πληροφόρηση των Ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά υπάρχει μία αδυναμία στις επαφές αυτές, διότι είδα τις διαβουλεύσεις και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προετών είχε οργανώσει ορισμένες διαβουλεύσεις, όχι πρόσφατα, λίγο πιο παλιά, σχετικά με το σύστημα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για την οργάνωση αυτού της εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και είχαν ε, λάβει 280 απαντήσεις και εγώ στη σελίδα μου του Facebook στην ε, Πολωνία οργάνωσα κάτι τέτοιο και έλαβα μόνο για την Πολωνία 450 απαντήσεις. Δέστε λοιπόν πώς λειτουργεί στο θέμα. Ε, μέσω του Facebook μόνο για την Πολωνία 450 απαντήσεις και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, Φόλης της ύλη και σε όλες τις χώρες 280 απαντήσεις. Δεν μου φαίνεται πολύ αξιόπιστο και καλύτερη συνεργασία, καλύτερη πληροφόρηση είναι ένα βασικό θέμα το οποίο προωθώ στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συζητητές και συζητητές για την λεπτομερέστατη δουλειά που έκαναν. Αυτό το θέμα το είχαμε ήδη συζητήσει, δηλαδή η συμμετοπρέτων κ. Ρόσφορντ παρουσίαζε την έκθεση για τους καταναλωτές. Ίσως θέλετε να προσθέσετε κάτι και από αυτού θα θέλαμε πρώτα να ακούσουμε την Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι μπορούν και όλοι οι σκιώδεις συγητές κάτι να μας πούν. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σφάμπ, ε, που είναι σκιώδης συγητής για την κύριο Μάιρ, κατόπιν ο Ρέκορ και μετά ο κύριος Ροσφόρ, Ρούντερ, Φόξ και Διόμερσερ. Αν υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν να μιλήσουν, να μας το πούν, να σηκώσουν το χέρι τους. Head, Hanslick, άλλοι. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα με την εντολή του συναδέλφου Hans Peter Mayer θέλω να εκφράσω τη δική του ή τις δικές μας απόψεις για την έκθεση του κυρίου Λουί Γκρέκ. Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Και ήδη με SMS έχω πει ότι με τις ουσιοδέστερες προτάσεις της εκθεσής του έχω πει στον κύριο Γκρέκο ότι τις δεχόμαστε και ως ΕΛΚΑ του ευχόμαστε κάθε καλό να αναρρώσει σύντομα και κάθε επιτυχία. Για την πρόταση αυτή έχει εδώ μια περιεκτική έκθεση που μας υποβάλλει και πολλές από αυτές τις τροπολογίες που έχει καταθέσει σίγουρα μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την προθεσμία 90 ημερών ως διορία που προτείνει και τις πιθανές εξαιρέσεις από πολλές πλευρές ζητήθηκε να μην υπάρξει προσδιορισμός προθεσμίας ή να υπάρχει ένα επαρκές χρονικό πλαίσιο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ένα σύστημα χωρίς διορίες και προθεσμίες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι λειτουργικό ένα σύστημα χωρίς προθεσμίες και ρυθμίσεις για διορίες και προθεσμίες. Ιδιαίτερα για τις διεργασίες των small claims δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς προθεσμίες. Γι' αυτό πολύ εξειδικευμένα και πολύ σύντομα θέλω να αναφερθώ στα σημεία εκείνα που θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Πρώτον, το θέμα της ολοκλήρωσης των ήδη υφισταμένων συστημάτων και ένταξή του σε αυτή την οδηγία επιδιαιτησίας. Δεύτερον, πώς θα διαμορφωθούν τα κόστη και οι δαπάνες με σωστό τρόπο. Τρίτον, το θέμα με ποιο τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κυρίας Ρώσα Τούν, δηλαδή στο πεδίο εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών δυνατοτήτων διαιτησία για τα εθνικά συστήματα, να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί, αν θα γίνει δεσμευτικού χαρακτήρα ή αν θα αναφέρονται κάποιοι στόχοι μόνο. Τέταρτον, το θέμα να δούμε αν θα επιτρέψουμε θέματα επιδιατησίας που θέλει να εντάσσονται ε, ε, καταναλωτές ή επιχειρηματίες ή αν θα υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα για τέτοιου είδους ανάγκες. Εδώ υπάρχουν και άλλα ίσονος, θέματα, ε, ίσονος ε, σπουδαιότητας θέματα. Αν μπορούν αυτά χωρίς γραφειοκρατική επιβάρυνση να διαμορφωθούν ίσως σε κάποια σημεία πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Το δεύτερο θέμα είναι οι συλλογικέ προσφυγές. Ο Hans Peter Mayer θέλει να επισημάνει ότι εδώ για τις συλλογικέ προσφυγές θα είναι ένα εξοδικαστικό σύστημα νομικά μη δεσμευτικό και τέλος και είναι το τελευταίο σημείο, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αυτοματοποιημένα δεσμευτικές αποφάσεις. Αποφασιστική σημασία δεσμευτικού χαρακτήρα είναι μια απόφαση δικαστηρίου, νομολογία δικαστηρίου. Τώρα, σύντομα για, αυτά τα, το, για το πρώτο από τα πέντε αυτά σημεία. Για το πρώτο, θεωρούμε ότι τα ήδη υφιστάμενα συστήματα που πιθανόν όσον αφορά την αμεροληψία, εσείς χρησιμοποίησατε τον όρο ανεξαρτησία. Δεν ξέρω αν είναι, θα είναι ανεξάρτητη αυτή η υπηρεσία, αλλά πρέπει να είναι αμερόληπτη. Πώς θα διασφαλίζεται η αμεροληψία. Έχουμε για λόγους κόστους ε, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται κάποιες ε, τροποποιήσεις ή αλλαγές. Δεύτερο σημείο, σημείο το κόστος. Στη σημερινή διατύπωση του Λουί Γκρέκ λέει, χωρίς κόστος ή τέλη συστήματα και σε εξαίρεση θα εισπράτεται κόστος ε, ή τέλος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εποφελές ε, όσον αφορά το κόστος. Πρέπει να είναι ισοδύναμο το αποτέλεσμα, να μην δημιουργείται υπερβολικό κόστος στα κράτη-μέλη και ο καταναλωτής να μπορεί να κατανοήσει ότι ένα τέτοιο σύστημα έχει πραγματικά την λειτουργία του και την σκοπιμότητά του. Πώς θα διαμορφώνεται αυτό ώστε να είναι θελκτικό για τους καταναλωτές δεν το έχουμε καθορίσει ακόμα. Δεν έχουμε κάποιες προτάσεις. Θα υποβληθούν όμως στη συνέχεια γιατί πρέπει να καλυφθεί αυτό. Για τις ε, διακρατικές, ε, διασυνοριακές τέτοιες ε, συμφωνίες προτείνεται να υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Αλλά όποιος πιστεύει ότι μια δεσμευτική τέτοια εισαγωγή σε διακρατικές περιπτώσεις για λόγους αρμοδιότητας δεν μπορεί να να διεκδικηθεί θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, σε σχέση με θέματα τριβών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Αυτό που θέλει να δούμε ο κύριος Σανς Πέτερ Μάιερ είναι να επιτρέψουμε ρητά και κατηγορηματικά ή επιχειρηματίες να μπορούν σε ε, έκτακτες περιπτώσεις να στρέφονται στην επιδιαιτησία και εκείνη. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να ρυθμιστεί υπό την ε, αιγίδα της Δανέζικης ε, Προεδρίας και γοργά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όχι μόνο για την ένταξη ODR και ADR αλλά να δούμε πώς και με την νομική επιτροπή θα προχωρήσουμε για μια ενισχυμένη συνεργασία με βάση το άρθρο 50 ώστε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η δυνατότητα μεταξύ συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Good. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το δούμε αργότερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα των corporation είναι εντάξει. Ο κύριος Ρέπο ε, είναι ο σκιώδης ηγητής ε, και δίνω το λόγο. Είχα την τιμή να ασχοληθώ ως σχεδόν εισηγητής ε, της ε, ομάδας ε, των Σοσιαλδημοκρατών με αυτό το θέμα. Είχα την ευκαιρία ως σχεδόν εισηγητής να ασχοληθώ από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να εκθέσω κάποια θέματα που μας απασχολούν. Πρώτον, εφιστούμε την προσοχή για το γεγονός ότι με τη σημερινή πρόταση το να έχουμε προθεσμίες ή διορίες που θα είναι υπερβολικά πιεστικές και σύντομες θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και δεν θα ήταν προ όφελο τη προστασία των καταναλωτών. Αν έχουμε πολύ πιεστικές τέτοιε προθεσμίες θα είμαστε πολύ βιαστικοί να υιοθετηθεί μια απόφαση γοργά και βιαστικά και με τη βιασύνη αυτή δεν θα διασφαλίζαμε το επαρκές πλαίσιο προστασίας καταναλωτών. Φυσικά κατανοώ το μέλημα, την ανησυχία να μην είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες αυτές οι προθεσμίες αλλά πρέπει να είναι επαρκή ώστε να διασφαλίζεται επαρκής κάλυψη των καταναλωτών. Θα ήθελα για το θέμα των μεταφράσεων να αναφέρω ότι η ποιότητα των μεταφράσεων είναι και αυτό ένα στοιχείο σημαντικό. Όταν έχουμε συμπιεσμένες προθεσμίες και η ποιότητα των μεταφράσεων μέσα σε αυτές τις συμπιεσμένες προθεσμίες, πιεστικές προθεσμίες ε, είναι ε, μη ικανοποιητική. Γι' αυτό θα ήθελα με περισσότερο εξειδικευμένα επιχειρήματα να μου εκθέσετε πώς θα προχωρήσουμε με τις μεταφράσεις σε τόσο πιεστικές ε, προθεσμίες. Η μόνη δυνατότητα που θα υπήρχε θα ήταν η αυτόματη μετάφραση, μια δυνατότητα αυτόματων μεταφράσεων. Αλλά τι μπορεί να γίνει. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά με τα δικά μας θεσμικά όργανα και διεθνή θεσμικά όργανα ε, δαπανώνται κονδύλια για τις μεταφράσεις και για τη διερμηνία λοιπόν τώρα για τους καταναλωτές. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε ένα σε επίπεδο ποιοτικό. Δεν πρέπει να μπορούμε να απαιτήσουμε να υπαρκούνται με μεταφράσεις ε, μη ικανοποιητικέ, πολύ βιαστικές ή στο γόνατο. Διότι όπως είπα αυτό δεν θα συνεισφέρει προς ε, την προστασία των καταναλωτών σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι στην οδηγία και στον κανονισμό για την ε, εναλλακτική επίλυση και διευθέτηση ε, μέσω του ηλεκτρονικού ε, των, των ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να έχουμε παρόμοιε προθεσμίε, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Με τη συνεργασία από πλευρά εισηγητού μπορούμε να προχωρήσουμε στη διευθέτηση αυτών των προβλημάτων. Εν πάση όμω περιπτώσει εδώ αυτό που θέλουμε είναι να προστατεύουμε πολύ πιο αποτελεσματικά του καταναλωτέ, ιδιαίτερα στι συναλλαγέ με το ηλεκτρονικό μέσο, το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Um, λοιπόν, ε, οι σχεδόν και για τις δύο προτάσεις από τις άλλες ομάδε, ξεκινώντας από τον κύριο Ροσφόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, είμαι σκιώδη ηγητή και για τις δύο εκθέσεις. Ξεκινάω με τι εναλλακτικέ του κυρίου Γκρέσ. Και εγώ του εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα και ήθελα να το συγχαρώ επειδή πράγματι η έκθεσή του είναι πολύ θετική και πολύ καλά συνταγμένη. Ξεκινώ λέγοντα ότι στα όσα υπενθύμισε η κυρία Γκέρχαρτ, συμφωνώ με το γεγονό ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή ε, των ADR στου καταναλωτέ. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό επί το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Τώρα έρχομαι στο πιο ευαίσθητο και λεπτό σημείο, επί το οποίο θα θέλαμε μια βελτίωση του κειμένου του κ. Γκρέσ. Αυτό έχει σχέση ε, με την πραγματική κατάσταση σε ορισμενα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ότι προ το παρόν υπάρχουν ε, μεσολαβητέ οι οποίοι ασχολούνται με μία μόνη επιχείρηση. Και τι κάνουμε σε μία οργάνωση γενικότερη μορφή. Δεν θα θέλαμε να κάνουμε τάμπουλα ράζα με τα όσα λειτουργούν καλά και με τα όσα δημιουργήθηκαν προτού οι μεσολαβητές μεταξύ επιχειρήσεων καταφθάσουν. Για μια χώρα όπως η δική μου, τη Γαλλία, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή εθνικοποιήθηκαν, ήταν πρώην μονοπόλια. Αυτό είναι λογικό, επειδή εκπροσωπείται πολύ αυτό, ο τομέας αυτός από μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Λοιπόν, θα ήθελα να βρεθεί μια, ένα συμβιβασμό μεταξύ των πολλών απαιτήσεων που έχουμε όσον αφορά την ανεξαρτησία που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι μεσολαβητές και, και από την άλλη πλευρά να διατηρήσουμε ε, την ύπαρξη μεσολαβητών σε μια πολύ πολύ μεγάλη επιχείρηση. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σύσταση ανεξαρτησίας όπως έγινε το 1998, αλλά ίσως να προτείνουμε πιθανόν και μια ξεχωριστή νομική επιβεβαίωση ε, της ε, ε, επιχείρησης όπου βρίσκεται, όπου λειτουργεί ο μεσολαβητής. Αυτό θα το δούμε με τον κύριο Γκρέσ, υπομορφή τροπολογιών τις προσεχείς ημέρες. Συμφωνώ με την επιθυμία εδώ συμφωνούμε, το είπε ο κύριος Σουάβ για το ΕΛΚ, συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση των καταναλωτών στις μορφές διαμεσολάβησης. Αυτό θα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο κρατών μελών, αφήνοντα όμω μεγάλη ευελιξία στην οργάνωση. Από την άλλη πλευρά όμω θα ήθελα, και ο κ. Άρμπο αναφέρθηκε σε αυτό που είπατε πρωτήτερα, δηλαδή αυτό το οποίο ε, φορούσα το άλλο καπέλο μου πριν, εισηγητή για το πρόγραμμα των καταναλωτών. Δεν είμαι πολύ σύμφωνο με την τροπολογία 33 που προβλέπει ότι το πρόγραμμα καταναλωτών θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει Νέε διαδικασίε εναλλακτική ρύθμιση των διαφορών. Νομίζω ότι ήδη δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο πρόγραμμα καταναλωτών. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάζεται στου οριζόμενου στόχου. Αυτό είναι ένα σημείο επί του οποίου δεν συμμερίζομαι την άποψη ε, του κυρίου Γκρέσο. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα. Προσωπικά συμφωνώ με την κυρία Τούν που λέει θα πρέπει να είναι το ίδιο χρονοδιάγραμμα και στι δύο περιπτώσει. Νομίζω ότι 90 ημέρε. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερα να είναι ημερολογιακές μέρες και όχι εργάσιμες ημέρες. Καλύτερα για τον καταναλωτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Συμφωνώ επίσης για το με την πρόταση του κύριου Γκρέσ, επειδή προτείνει λογικά πράγματα όταν λέει ότι η εναλλακτική μορφή ε, πύλης των διαφορών θα πρέπει να φαίνεται ε, ευδιάκριτα στα έγγραφα. Δηλαδή να είναι με ένα μεγάλο διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ζητώντα δηλαδή αυτό να αναγράφεται ε, σε κάθε τιμολόγηση, σε κάθε απόδειξη. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι νομίζω ότι είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί η ανασταλτική πτυχή της προσφυγής ή των εναλλακτικών μεθόδων για επίλυση των διαφορών. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα σταλτικό χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί κανείς να εφεσιβάλει ε, τις περιπτώσεις που έχουν καθαρά δικαστική μορφή. Τώρα, για την έκθεση της κυρίας Τούν. Τον ευχαριστώ επίσης για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που έκανε. Απλώς και μόνο θα ήθελα να σας πω ότι από τη στιγμή που η πλατφόρμα των ODR είναι μάλλον πλατφόρμα τελειοποίησης παρά επίλυσης των διαφορών, πιστεύω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ότι στις μορφές online να υπάρχει και η δυνατότητα ε, να καταλήξει κανείς το ίδιο αποτέλεσμα ε, με το αποτέλεσμα που θα είχαμε ήταν διαφορέ offline. Δηλαδή, αν μια διαφορά είναι offline, θα μπορούσαμε πάλι να στραφούμε σε αυτή την πλατφόρμα τελειοποίηση και να ακολουθήσουμε τις κανονικές διαδικασίες. Είναι μια μορφή dispatching. Τώρα, για τα όσα είπε η κυρία Τούν, ότι δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει ήδη να ενσωματωθούν ε, στις σελίδες που γνωρίζει ο καταναλωτής, οι ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ ε, να μην γίνουν αυτές οι ιστοσελίδες ε, κάτι που τα περιλαμβάνει όλα, που δημιουργεί σύγχυση και τελικά ο καταναλωτής να μην βρίσκει το δρόμο του, όπως λέμε, και να μην βρίσκει τις σωστές σελίδες, τις σωστές προσβάσεις. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ακόμα κι αν είναι online, η επίλυση των διαφορών δεν θα γίνει καταρχήν από τους πολύ ηλικιωμένου καταναλωτές και γι' αυτό η ευελιξία τους να περιπλανώνται στον παγκόσμιο ιστό ε, έχει σχέση με την γενεά στην οποία ανήκουμε. Γι' αυτό όλες οι πλατφόρμες που έχουν σχέση με τα ODR, ε, συμφωνεί η κυρία Τούν φαντάζομαι, θα πρέπει να είναι φιλικές προς τον χρήστη, οι πληροφορίες να είναι σαφείς, κατανοητές, θα πρέπει να προβλέψουμε τις ερωτήσεις που θα κάνει ο καταναλωτής και να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που δεν έχουν ε, τόση ευχέρεια με τη χρήση των υπολογιστών. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να σας κάνω. Τε, τελειώνοντας, δεν ξέρω αν συμφωνώ απόλυτα με την σημειολογική παρατήρηση της κυρίας Τόπου. Λέει, ε, facilitator ή σύμβουλος διευκολυντής, δηλαδή νομίζω ότι οι εναλλακτικές μορφές επίλυση των διαφορών είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συμβουλή ή γνώμη. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο επιλύει τη διαφορά δεν ξέρω αν είναι γλωσσικό το πρόβλημά μου και ανάλογα με τις μεταφράσεις μπορεί κανείς πιο εύκολα να βρει μια λέξη για τον σύμβουλο, αλλά για έναν Γάλλο σύμβουλος περιορίζει κάπως το εύρος, τη σημασία. Ενός facilitator είναι ένας όρος που λέει ότι θα διευκολύνει την κατάσταση. Ε, είναι κάτι πιο ισχυρό από το απλό γεγονός ότι δίνει κανείς τη συμβουλή του. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές διότι ε, δεν τα ξέρω όλα αλλά θα ξεκινήσω με το ODR όπου πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να εξισωθούν οι προθεσμίες για τα ODR και ADR και οι 90 ημέρες μου φαίνονται σωστές και ε, δεν ε, ε, βλέπω ότι και το Υπουργείο μας προτείνει τις 90 ημέρες ε, που θεωρώ ρεαλιστικό. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά είναι σωστό να μπουν σε μία τελευταία σελίδα της ηλεκτρονικής ε, ιστοσελίδας ε, του ε, Europe διότι όπως ο κύριος Ροσφόρ πιστεύω ότι δεν θα βρίσκουν άκρη οι καταναλωτές δηλαδή αυτοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο δεν θα, δεν θα καταφέρουν να προσανατολιστούν Κατά τα άλλα όμως συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Τούν και τη στηρίζω και έχω ορισμένες παρατηρήσεις δηλαδή ε, πρέπει να περιοριστούμε ε, ε, εις τα μέτρα τα οποία υπάρχουν υπάρχουν ορισμένα τα οποία δεν αναφέρονται εδώ και εγώ έχω ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την ενημέρωση. Πιστεύω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούμε και να τα αναδιατυπώσουμε και σήμερα το πρωί για το breakfast υπήρχαν ορισμένες πληροφορίες, δηλαδή πιστεύω ότι η υπερβολική πληροφόρηση τρομάζει τον καταναλωτή, πιο βασικό είναι να περιοριστούμε στα ουσιώδη. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι όλα και ε, γενικώ αυτά είχα να σας πω. Πολύ καλά. Βλέπω ότι προσθέτεται πράγματα και αξία. Κύριε Σπόξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα για το ADR. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρέγ για την εργασία και την κυρία Γκέπαρτ που έκανε την παρουσίαση. Δέχομαι πολλές από τις προτινόμενες αλλαγές και συμφωνώ με πολλούς από τους στόχους του εισηγητή αύξηση της κάλυψη EDR και της προσβασιμότητας του EDR. Οι εμπορευόμενοι καταναλωτές να γνωρίζουν ποιο είναι το ADR και τα ωφέλη. Ε, γενική ελάχιστη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του ADR για να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα. Αλλά επίσης ε, τον σεβασμό των εθνικών προγραμμάτων ε, που έχουν μεγάλη προστασία των καταναλωτών και λαμβάνουν υπόψη τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας και κυρίω αναφέρουμε στο γαλλικό σύστημα το οποίο μας υπογράμμισε ο κύριος Ροσφόρ. Αν λειτουργεί για τη Γαλλία, γιατί εμείς να θέλουμε να το αλλάξουμε. Συμφωνώ με τη βελτίωση της προσβασιμότητας ε, από όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι ως, να έχει ως τίμημα την καταστροφή των υπαρχόντων συστημάτων όπως της χώρας μου. Θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά και όχι να τα αποκαταστήσουν, κυρίως εκείνα που έχουν διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Με χαρά βλέπω ότι ο εισηγητής αποκλεί ε, τις, ε, των επιχειρήσεων να καταθέτουν αυτά τα παράπονα. Ένα από τα αντικείμενα είναι να αποκαταστήσουμε την ανισορροπία ισχύω μεταξύ των μερών και δεν θέλουμε οι καταναλωτές να μην ακολουθούν αυτόν τον σκοπό. Συμφωνώ να έχουμε κανόνες, διαδικασίες που επιτρέπουν στις μονάδες ADR να επιλύουν τις διαφορές ο εισηγητής αναγνωρίζει την ανάγκη ε, ευελιξίας, κυρίως για τις περίπλοκες περιπτώσεις. Αναφέρομαι στις διαφορές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που απαιτούν περισσότερες από 90 μέρες. Για να έχουμε τα μέγιστα ωφέλη από την πρόταση, θα ήθελα να προσθέσω ορισμένε ακόμα τροπολογίες προκειμένου το ADR να είναι ε, ε, δωρεάν για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους. Το ADR να είναι πιο ελκυστικό για τα δικαστήρια και να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες οι οποίες θα πρέπει να περιορίζουν ορισμένες αξιώσεις. Νομίζω θα πρέπει η βιομηχανία να το χρηματοδοτήσει. Δεν όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δύσκολες εποχές λιτότητας να πρέπει να πούν στα κράτη-μέλη ε, εσείς θα, ναι, δεν πρέπει, να το πούν στα κράτη-μέλη δεν πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής αλλά ούτε να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα, κράτη θα πληρώσουν. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ευελιξία σχετικά με τις μορφές των EDR. Ακόμα και η δυνατότητα της χώρας να αναθέσει ένα, ένα σχήμα ε, σε ένα τομέα, όπως το χρηματοπιστωτικό. Μετά από τα όσα είπε ο κ. Ροσφόρ, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία ε, σε εκείνο το οποίο θεωρούμε ανεξάρτητο. Αυτό είναι το πιο ευαίσθητο πολιτικά θέμα σε αυτό το φάκελο. Και μετά από την επιστολή των τεσσάρων κρατών μελών, θα ήθελα να παρατηρήσω τον κύριο Γκρέκ και του άλλου και όλους τους να βρουν μια, ένα αποδεκτό συμβιβασμό για να μην διαλύσουμε τα υπάρχοντα συστήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί σωστά. Θα ήθελα τώρα, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω για τα ODR Ευχαριστώ την κυρία Τούν για το έργο που επιτέλεσε. Ε, νομίζω ότι μας είπε ότι υπήρχαν ορισμένε αδυναμίες μεταξύ της Επιτροπής ε, και των καταναλωτών. Ε, νομίζω ότι εάν η κυρία Τούν είχε 400 απαντήσεις στο Facebook μόνο στην Πολωνία ε, σε διαστολή με τα 450 της Επιτροπής. Πώς μπορεί να το λέει αυτό. Ε, πολλές τροπολογίες ε, της κυρίας Τούν είναι καλές και προσθέτουν κάτι στην πρόταση της Επιτροπής. Αλλά ε, υπογραμμίζω την ανάγκη αποφυγής των επικαλύψεων και το, το πιο προφανές παράδειγμα είναι το γεγονό ότι τα αρχικά παράπονα μπορούν να γίνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της κοινότητας. Πρέπει να καταστεί σαφές από την αρχή ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να περιμένει ότι η μονάδα DR θα λειτουργεί στην ε, γλώσσα του καταναλωτή. Αυτό απλώς και μόνο είναι αδύνατον και θα επέβαλε μεγάλο βάρος ε, στις μονάδες ε, DR στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι η λύση default είναι εκείνη, εναλλακτική λύση δηλαδή, είναι εκείνη που σας δίνεται σε αυτό το έγγραφο που λέει ότι η λύση default θα πρέπει ε, να είναι η λύση, δηλαδή ε, η μορφή του EDR θα είναι ε, στη γλώσσα της σύμβασης. Εάν μπορεί λοιπόν να συναυθεί σύμβαση σε μία αλφα γλώσσα, τότε μπορεί κανείς ε, να συναγάγει ότι το άτομο που θέλει να αναγνώσει το ADR θα καταλαβαίνει τη γλώσσα. Αυτή είναι μια θέση default, ώστε ε, και οι επιχειρήσει ε, Και... Οι επιχειρήσει λοιπόν μπορεί να είναι διατεθειμένε να το χρησιμοποιήσουν ή να υποχρεωθούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό σύστημα. Πρόεδρε, θα ήθελα επίση να αναφερθώ σε ορισμένε τροπολογίε. Δεν συμφωνώ με την τροπολογία 21, η οποία ορίζει ότι η διαδικασία είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν αυτή η διαδικασία. Κάποιος πληρώνει, πιθανόν ο φορολογούμενος. Νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ότι κάτι είναι δωρεάν. Δωρεάν κάποιος πληρώνει. Ε, αν δεν το πληρώνει η επιχείρηση και ο καταναλωτής, το πληρώνει ο φορολογούμενος. Οι τροπολογίες 29 και 30 προσθέτουν δαπάνες και βάρος στο σύστημα όσον αφορά την πύλη. Και η τροπολογία 33, κατά την άποψή μου, ε, δεν είναι σωστή. Δεδομένου ότι διευκολύνει τους καταναλωτές να δώσουν ε, αντικειμενικές απόψεις για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μονάδων ADR. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με άκουσαν και προσβλέπω στη συνεργασία με, τον κύριο και, με την κυρία Τόν και τον κύριο Γκρέγκ. Ευχαριστώ για την πολύ σαφή τοποθέτησή σας και είναι προφανές ότι οι συγητές και οι ισχυώδεις συγητές εργάζονται χέρι με χέρι το οποίο είναι βασικό. Η κυρία Χέντ ήθελε να μιλήσει, κάποιος άλλος. Ε, ξέχασα τον κύριο Ντιόν. Με συγχωρείτε, ο κύριος Ντυρό ήρθε καθυστερημένος, έχουμε όμως ακόμη έναν ε, σκιώδη συγγητή. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, θέλω να σας πω ότι θα περιορίσω τα σχόλιά μου εις τα ADR διότι Βλέπω ότι δεν έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις. Ευχαριστώ τον Λουί Γκρέχ για, όλες, ε, για την παρουσίασή του. Και όσον αφορά τη θέση μου σαν σκιώδη συγητή, πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε και συμφωνώ για αυτό το οποίο ελέγχθη, ότι χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία επί του θέματος αυτού, και ε, δεν πρέπει να γίνεται η κατάσταση πιο δύσκολη από ό,τι είναι απαραίτητο. Ε, υπάρχει ένα ποσοστό αυτορύθμισης, το σύστημα λειτουργεί κανονικά, δεν πρέπει να δυσχεράνουμε την κατάσταση και να μην ε, ε, θέτουμε σε κίνδυνο ένα εύρυθμο σύστημα μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από πλευράς οικονομικής πιστεύω ότι είναι απλό να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν διάφορα σήμερα, αλλά δεν είναι πάντοτε προφανές να γίνει κάτι τέτοιο, διότι από τη μία πλευρά λέμε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε πόρους και από την άλλη πλευρά ζητούμε από τα κράτη-μέλη κάνουν ένα σωρό πράγματα τα οποία ε, είναι δαπανηρά, χρειάζονται χρήματα. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη να ε, χρηματοδοτήσουν αυτά, διότι υπάρχουν συστήματα ήδη λειτουργία, τα οποία λειτουργούν ε, ικανοποιητικά όσον αφορά την την ανεξαρτησία πρέπει να είμαστε ε, ευέλικτοι όπως σας είπα και να σκεφτόμαστε ε, και το οικονομικό θέμα. Δηλαδή να υπάρξει μία πρακτική διασύνδεση με την ε, εμπλεκόμενη βιομηχανία και να καλύπτουμε τους καταναλωτές. Συμφωνώ επίσης ότι ε, ε, θα, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή περισσότερο και όχι τόσο πολύ ε, να καλύψουμε τα παράπονα των επιχειρήσεων και όσον αφορά τις 90 μέρες προθεσμία για περίπλοκα θέματα Φαντάζομαι ότι υπάρχει μία μία αλλαγή. Θα προτιμούσα λοιπόν αυτό το οποίο προτείνει εδώ η Επιτροπή και να διατηρηθεί. Η οργανώσεις καταναλωτών είπαν ότι θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε νομική, νομικές συμβουλές αλλά πιστεύω ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η μία πλευρά θα πρέπει να αποκλείεται από την νομική έμπειρη γνώμη και από προσφυγή στα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Head σύντομα παρακαλώ, γιατί θα ήθελα να ολοκληρώσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση, την έκθεση Λουίς Γκρέκ, σε αυτήν αναφέρομαι. Ο συνάδελφος ευφιέστατα προτείνει τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τους καταναλωτές με τέτοιες προσφυγές και όχι με τις επιχειρήσεις. Ε? Υπάρχουν άλλα φόρα για την επιδιαιτησία όσον αφορά θέματα επιχειρήσεων. Δεν θα ήταν καλό να αναμειχθούν οι επιχειρήσεις σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα επιδιαιτησίας καταναλωτών. Πέρα από αυτό, τα αρμόδια όργανα τα οποία καλύπτονται από αυτή την οδηγία από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρονται σε σχέση με το άρθρο 17β να το συζητήσουμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, πώς μπορούν να διαθέτουν πληροφορίες σε σχέση με αυτές ε, τις υπηρεσίες. Χρειάζονται οι καταναλωτές τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες προτού συνάψουν ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση. Δεν πρέπει όμως να δημιουργούν προσκόμματα και εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το βλέπει το θέμα της διάθεσης, διαθεσιμότητας ε, πληροφοριών και ενημέρωσης όσον αφορά τι ε, μικρέ επιχειρήσει σε σχέση με την πρόταση. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Κριστίνα Ρούσο να τοποθετηθεί. Σύντομα σχόλια και μετά από την κυρία Γκέπχαρτ και την κυρία Τόν και θα ολοκληρώσουμε μετά και θα κλείσουμε αυτόν τον πρώτο γύρο συζητήσεων. Α, και από πλευρά σας εσεί θέλετε να παρέμβατε. Συγγνώμη που δεν σας είδα. Δεν είχαμε το όνομά σα στον κατάλογο. Δεν βρισκόταν στο δικό μου κατάλογο το όνομά σα τουλάχιστον. Η κυρία Χάνσλε πρώτη λοιπόν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είχα στραφεί στη γραμματεία για την παρέμβασή μου, αλλά δεν πειράζει. Σύντομα θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές όμως για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν, πρέπει να πω. Το ODR και το ADR θα έπρεπε τις ε, επιδιατησίες ως μηχανισμοί να τις ρυθμίζουν αποτελεσματικά. Άκουσα όλες τις προτάσεις που έγιναν, δεν μπορώ όμως να συμφωνήσω με όλα. Με ανησυχεί ένα θέμα, το μέλημα το οποίο έχω σε σχέση με αυτά που είπε η συνάδελφος εκπροσωπώντας τον κύριο Γκρέκ όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα να το ξανασκεφτούμε θα ήθελα. Και θα ήθελα να μου πείτε κάτι να μου το αποσαφηνίσετε. Το ανέφερε η κυρία Τούν, το ανέφερε και ο συνάδελφος των σοσιαλδημοκρατών. Αυτή η μηχανική μετάφραση, η αυτοματοποιημένη μετάφραση όσον αφορά τέτοιες μεταφράσεις μέσω μηχανών. Όταν τροφοδοτούμε αυτές τις μηχανές με ένα κείμενο που θέλουμε να μεταφραστεί. Είχαμε και ένα παράδειγμα από τα πολωνικά στα αγγλικά. Μεταφράστηκε ο μιλητής ως μεγάφωνο, δηλαδή speaker σε loud speaker. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε, μπορεί αυτή η μετάφραση μηχανικά, αυτοματοποιημένα να λειτουργήσει σωστά. Τι γίνεται με τις λειτουργικές δυνατότητες τέτοιων μεταφράσεων, μηχανικά ή αυτοματοποιημένα είναι επιτυχής, ε, υπόσχονται πολλά. Ίσως ε, αυτό το θέμα θα πρέπει στην ε, γλώσσα σύμβασης, ολοκλήρωση ολοκλήρωσης της σύμβασης να βασιστούμε ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή το συμβόλαιο το οποίο συνάπτεται ε, στη γλώσσα αυτού θα πρέπει να ε, διεξάγεται η επιδιατησία Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το είπε και η κυρία Τούν πιο πριν. Και τελευταίο σημείο ως παρατήρηση. Θα έλεγα καλό θα ήταν αν θα μπορούσαν οι καταναλωτές να γνωρίζουν όλα αυτά τα στοιχεία, διότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν και δεν ε, ποια είναι τα δικαιώματά τους και δεν ξέρουν από πού πρέπει να πληροφορηθούν και να πάρουν αυτές τις πληροφορίες που είναι και σημαντικές κιόλα. Όλα αυτά λοιπόν σε μια ιστοσελίδα, σε μια ιστοπύλη Europortal μπορούν να καλυφθούν έτσι. Γιατί ίσως αυτό θα ήταν μια δυνατότητα. Μια δυνατότητα να έχουμε μια κοινή πρόσβαση ODR, ADR για να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ ολοκλήρω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ρούσο, παρακαλώ. Με συγχωρείτε που σας έκανα να περιμένετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όσο δυνατόν συντομότερη, επειδή δεν υπάρχει χρόνος. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας για τη δουλειά που κάνατε, κυρίως την εισηγήτρια την κυρία Τούν και τον κύριο Γκρέκ και θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να πείτε ε, τις ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση στον εισηγητή. το βασικό, τα βασικά θέματα παρουσιάστηκαν από την Γεια Γκέρμπερ, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας βρίσκουν σύμφωνος, κυρίως όσον αφορά τα τρία σημεία για να καλύψουμε τα κενά ε, η τομεακή και γραφική κάλυψη, η ποιότητα και οι ανάγκες για πληροφόρηση. Τώρα, οι ανάγκες για πληροφόρηση, που είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε και από άλλα αξιό τη Μαμέλ, τον κύριο Ροσφόρ, κύριε Χέτ, θα προτιμούσαμε να διατηρηθούν οι πληροφορίες επάνω σε αποδείξεις και τα τιμολόγια ε, πρέπει να βρεθεί μια λύση για να αποκλειστούν οι μικρές επιχειρήσεις. Ίσως στην πρότασή μα θα έπρεπε να πούμε μεγαλύτερη σαφήνεια ότι αυτές οι πληροφορίε θα πρέπει να γίνουν για να βοηθήσουν την EDR και όχι για να παρεμβαίνουν στη λειτουργία του OEDR. Ε, Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να εξετάσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα αλλά είμαστε ευγνώμονε ε, στον κύριο Γκρέγκ επειδή αυτό είναι από τα σημεία επί του οποίου και το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, έχουν επιμείνει. Επίσης θα ήθελα να ότι πρέπει να καλύψουμε στο ODR και τα εσωτερικά θέματα και τα διασυνοριακά και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση της Κυριαρτουν για το ODR και βλέπω ε, λογική να επεκτείνουμε την πλατφόρμα και στα διασυνοριακά και στα εσωτερικά, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσουμε, ανταποκριθούμε καλύτερα ε, στις ε, πολιτικές απαιτήσεις της ψηφιακής ατζέντα. Ένα θέμα που θα συζητήσετε σήμερα το απόγευμα. Σκεφτήκαμε ότι κάποια άλλη στιγμή θα το συζητούσαμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά είμαι λίγο διστακτική τα όσα είπε ο κύριος Ροσφόρ για την επέκταση της πλατφόρμας στις περιπτώσεις offline. Ίσως για το γεγονός ότι αυτό θα είναι ένα βάρος για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις, επειδή αυτό θα σημαίνει ότι σε όλες τις συναλλαγές online ο, ε, το άτομο θα πρέπει να αναφέρει στον καταναλωτή την ιστοσελίδα του, ε, την ε, διεύθυνσή του για να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα. Λοιπόν, εδώ δεν συμφωνώ. Ένα άλλο πολύ λεπτό θέμα, οι δικλείδες ασφαλείας και ανεξαρτησία. Ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία υπόθηκαν. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μεγάλες δικλείδες ασφαλείας για να είναι ανεξάρτητες οι μονάδες ADR. Και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ε, της κατάστασης από πλευράς Κοινοβουλίου. Τώρα, για τα θέματα της κυρίας Τούν, συμφωνούμε την πρόθεσή σας να απλουστεύσετε το σύστημα, να το καταστήσετε πιο προσβάσιμο στους καταναλωτές και να το καταστήσετε όσο δυνατόν αποτελεσματικότερο. Τώρα, ως προς τη θέση με το Europe, όπως ε, αυτό αναφέρθηκε και από άλλους, πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, πύλη όσο το δυνατόν περισσότερο, αποφεύγοντα όμως να δημιουργηθεί ένα επιπλέον στάδιο που θα πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτή. Γιατί αυτή η, η, πλατφόρμα ω αντικείμενο έχει την άμεση πρόσβαση από τον καταναλωτή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη συνοχή και εύκολη πρόσβαση από του καταναλωτέ. Για τι προθεσμίε σημειώνουμε τα όσα υπόθηκαν θα προτιμούσαμε μια κοντύτερη προθεσμία για το ODR, αλλά μπορούμε να δεχθούμε και τις 90 μέρες και για τα δύο. Τώρα για τις δεσμευτικές ή δεσμευτικές αποφάσεις για το EDR, η πρόταση της Επιτροπής το αφήνει ανοιχτό. Και ε, θα ήθελα να απαντήσω τώρα στην κυρία το τον κύριο Σφόξχολ, για το θέμα της ευελιξίας. Εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε στα υπάρχοντα στα κράτη-μέλη να καλύψουμε τα κενά, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα υπάρχοντα EDR και τα καινούργια EDR να εξασφαλίζουν ε, ότι θα, υπάρχουν, υπάρχει συμμόρφωση σε ελάχιστα κριτήρια ποιότητας. Επίσης, ε, πρέπει να, να συμφωνήσουμε στους ε, κανόνες. Ο κ. Φόξ αναφέρθηκε για τη γλώσσα των συμβάσεων και για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Συμφωνώ με την πρότασή σας και έρχομαι τώρα στο μεταφραστικό σύστημα. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μεταφραστικό μηχάνημα το οποίο δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό όσο περιμέναμε, αλλά η Επιτροπή διαμορφώνει ένα νέο μεταφραστικό μηχάνημα το οποίο θα υποστηρίζεται και από ανθρώπους, πραγματικούς ανθρώπους. Και ελπίζουμε ότι αυτό το μεταφραστικό μηχάνημα, η μηχανή, θα ανταποκριθεί ε, όσο δυνατόν σε απαιτήσει τη πλατφόρμα ODR. Επειδή δεν υπάρχει άλλο χρόνο, θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να κάλυψα τα πιο βασικά σημεία και, εν πάση περιπτώσει, είμαι στη διάθεσή σα για περαιτέρω ερωτήσει ε, επιδημερούς βάσεως. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ του διερμηνείς που έμειναν λίγο παραπάνω. Οι συγητές. Δεν έχουμε χρόνο για καταληκτικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι οι παρουσιάσεις που κάνετε ήταν πολύ καλές. Γι' αυτό θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τις, προθε... για τις τροπολογίες 21 Μαΐου 12 το μεσημέρι, εξετάση ε, τροπολογιών 21 Ιουνίου, συμβιβασμό 1 Ιουλίου, ψηφοφορία 10 Ιουλίου. Ευχαριστώ όλους για ε, τη θαυμάσια δουλειά που έκαναν μαζί ε, που αποδεικνύεται από την ποιότητα και τις λεπτομέρειες που ακούσαμε σήμερα και ευχαριστούμε επίσης την εκπρόσωπο της Επιτροπής που μας βοήθησε. Ε, ολοκληρώσαμε τις πρωινές μας εργασίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 το απόγευμα ακριβώς η κυρία Κρούς θα είναι εδώ για να μας μιλήσει για την ψηφιακή ατζέντα. Σας ελπίζω ως πρόεδρος της ομάδας μας για τα ψηφιακά θέματα και στις 4 θα ψηφίσουμε την έκθεση κ. Γκέφ Χάρσε, την πρόσβαση ε, των, στις βασικές υπηρεσίες. Φροντίστε να είσαστε εδώ για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη.